Eh, Καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. Θα αρχίσουμε αμέσως. Καλημέρα σας. Σας ε, καλωσορίζω στο σημερινό σεμινάριο. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αφρό προσέλευση. Δείχνετε τη δέσμευσή σας και θα συμβάλλουμε στην ε, κοινοτική στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους ιδιαίτερους τους προσκεκλημένους μας. Θα σας τους ε, παρουσιάσω όταν έρθει η ώρα να παρέμβουν. Κύριε Μπιλίντα Χφάη, καλώς ορίσατε. Είστε Γενική Διευθύντρια για τα θέματα ισότητας ε, των δύο φύλων. Ελπίζω ότι θα έχουμε χρόνο για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις όλων των παρισταμένων. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Σήμερα θα συζητήσουμε τις ανάγκες, ε, τα νέα εργαλεία που χρειαζόμαστε, ούτως ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική στρατηγική για την προάσπιση της ισότητας των δύο φύλων. Πέραν από τους προσκεκλημένους έχουμε την εισηγήτριά μας για την αντίστοιχη έκθεση, η κυρία Ήλντα Φιγκρέιντο. Εισαγωγικώς θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμά μας. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή ως προς το χρόνο αγόρευσης. Δείξτε λίγη αλληλεγγύη για να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις γίνεται. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή, ξαναλέω, με το χρόνο αγόρευσης. Θα αρχίσουμε με την ε, παρουσίαση της κυρίας Φιγκυρέιντο. Πέντε λεπτά κυρία Φιγκυρέιντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Ομίγυρη και τους προσκεκλημένους μας που δέχτηκαν να έρθουν να συμμετάσχουν στην σημερινή ακρόαση. Η συμβολή σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα θέλαμε κυρίως να μάθουμε ποια είναι η άποψή σας ως προς την εφαρμογή των μέτρων που έχουν αναλυφθεί σε επίπεδο ένωσης αλλά και σε κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος να γνωρίσουμε την άποψή σας για μια νέα στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων, την ισότητα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες για την κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης και των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η ανισότητα που σημειώνεται θα πρέπει να καταργηθεί μέσα από την κοινωνική πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση ως προς τα δικαιώματα όλης, όλων των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι το έτος που μόλις ξεκίνησε με μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά της και την ε, υπεσχημένη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διαρκέσει έως το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θέλουμε να διερευνήσουμε με ποιο τρόπο θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα στρατηγική για την ε, ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Δεδομένου του ότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι εξαιρετικά σοβαρή για τις γυναίκες. Είναι η εκατοστή επέτειος ε, της πρώτης ημέρας των γυναικών, η επέτειος των 15 ετών της ε, πλατφόρμας του Πεκίνου, Έχουμε τα στατιστικά δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούμε ποια είναι η καθημερινότητα των γυναικών και διαπιστώνουμε πως η ανεργία των γυναικών ανέρχεται σε λίγα ανησυχητικά ποσοστά. Η ένδυα που αγγίζει 85 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα γυναικείο πρόσωπο και οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν πληγεί περισσότερο από όλους από τη φτώχεια είναι αυξημένη η ανεργία και ε, είναι επισφαλής και κακώς αμοιβόμενες οι θέσεις εργασίας που έχουν. Υπάρχουν ακόμη ανισότητες ως προς τους μισθούς παρά τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί εδώ και 30 χρόνια και πλέον. Υπάρχουν επίσης δυσκολίες στην πρόσβαση στις ε, δημόσιες υπηρεσίες, στις πρόσβασεις σε ποιοτικέ υπηρεσίες για την περίθαλψη των παιδιών, για την περίθαλψη των ηλικιωμένων και ε, βαρύνονται οι γυναίκες ε, με περισσότερα καθήκοντα σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή ως προς τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Άρα χρειάζεται μία νέα στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη αυτήν την πραγματικότητα. Χρειάζονται μέτρα κρατικής παρέμβασης, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται και μία νέα νοοτροπία και πολιτικές προώθησης της ισότητας των δύο φύλων, ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γνωρίζουμε πως προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νέα στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων στα μέσα του έτος. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκπόνηση αυτής της στρατηγικής. Με και δρομολογούμε αυτές, αυτή τη διαδικασία με τη σημερινή ακρόαση και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με την έκθεση που θα εκπονήσει η Επιτροπή μας. Θα λάβουμε υπόψη τη συμβολή σας και ε, να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να μας αποστείλετε οποιαδήποτε στιγμή γραπτές παρεμβάσεις. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα από αυτές τις εργασίες που διοργανώνουμε. Όπως είπε η Πρόεδρός μας ήδη, θα έχουμε δύο πάνελ συζητήσεων. Το ένα για τις στόχους και τις προτεραιότητες για μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των Φίλων και μια άλλη ομάδα συζήτηση, ένα άλλο πάνελ για τα μέσα και τα εργαλεία για μια αποτελεσματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας. Ε, πέραν από τις ομιλήτριες που θα ακούσουμε, θα κάνουμε συζήτηση στην Επιτροπή μας μετά από τις πρώτες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Φιγκυρέντο. Καλωσορίζω την πρώτη προσκεκλημένη μας είναι η καθηγήτρια Σίλβια Ουάλμπι και είναι πρόεδρος σε θέματα ερευνών για τα δύο φύλλα στην UNESCO αλλά και στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ. Καλώς ορίσατε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε τις εξελίξει της στρατηγική ε, για την ισότητα των διαφύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την καλύτερη στρατηγική για την ισότητα των διαφύλων στον κόσμο. And it could be better. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και καλύτερη. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Θα συζητήσουμε λοιπόν κάποιου τρόπους με τους οποίου μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Ο οδικός χάρτη έχει σωστά παραθέσει πολλές από τις προκλήσεις. Υπάρχει ένα ερώτημα για το κατά πόσο τα προβλήματα αυτά έχουν λυθεί. Υπήρχε επίση ένα ερώτημα για την οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κλείσει το κενό που υπάρχει στις, στο μισθολογικό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης, συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακής ζωής. Πολύ λίγες χώρες έχουν επιτύχει τους ε, στόχους της Βαρκελόνης για την φροντίδα των παιδιών και σε πολλές χώρες δεν ξέρουν καν οι πολίτες ότι υπάρχουν τέτοιοι στόχοι. Η ε, ίση ε, εκπροσώπηση στην λήψη αποφάσεων. Φυσικά υπάρχει αυτό όμως στο Κοινοβούλιο, σε οικονομικούς κύκλους, σε ανώτερα κλιμάκια λήψη αποφάσεων. Επίσης, ε, ε, βία εναντίον των γυναικών. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά έχουμε ξεκινήσει να το λύνουμε. Απάλληψη όλων των στερεοτύπων που αφορούν τα φύλλα. Έχουμε επιτύχει στον τομέα της εκπαίδευσης. Αλλά ίσως να μην έχουμε επιτύχει στα ΜΜΕ και στην απασχόληση. Η πρόθεση των εξωτερικών πολιτικών σε σχέση με τα δύο φύλλα. Έχουν υπάρξει πολλές πρόοδοι εδώ, αλλά δεν, το, δεν τις γνωρίζουν πολύ. Και αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τομεί, σημαντικοί τομεί, στου οποίου μπορούμε να δράσουμε και τα προβλήματα των οποίων δεν έχουν ακόμη λυθεί. Υπάρχουν δύο αναδυόμενα θέματα, τα οποία είναι χρήσιμα για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Καταρχήν, τα δύο φύλλα και η οικονομική κρίση. Και λέγοντα αυτό δεν εννοώ την άνηση, ε, τις επιπτώσεις που έχει η κρίση στις γυναίκες, αλλά πώς οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αποτέλεσε ε, μία από τις αιτίες για την ε, οικονομική κρίση. Είναι λοιπόν ώρα να διορθώσουμε την έλλειψη αυτή των γυναικών στις οικονομικές αποφάσεις και να ενισχύσουμε την ε, ίση εκπροσώπηση στην λήψη αποφάσεων και στους ε, οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αναδιαρθώνοντας τους ε, οργανισμούς αυτούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε μια ακόμη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτή είναι η χρονική στιγμή η σωστή και αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε για την αναδιάρθρωση αυτών των οργανισμών δυνάμει των κατευθυντηρίων γραμμών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην λήψη αποφάσεων. Επίσης, έχουμε δεσμευθεί σε ό,τι αφορά το gender budgeting στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το εφαρμόσουμε πολύ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την, πολιτικέ. τις πολιτικές. Πολιτικές που έχουν προκύψει σε σχέση με την οικονομική κρίση. Έχουμε δει κάποιες πολιτικές που προσπάθησαν να ενισχύσουν την οικονομία και πολλά από τα κονδύλια αυτά κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της απασχόλησης, όπου οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται πλήρως. Τώρα περιμένουμε μεγάλη, ε, μεγάλες ε, μειώσεις των κρατών, από τα κράτη-μέλη, μεγάλες μειώσεις στους προπολογισμού και ξέρουμε ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι τομείς όπου ε, δεν προσωπούνται ισότιμα οι γυναίκες. Οπότε πρέπει αυτό να το δούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι ένα καυτό θέμα σε αυτή τη φάση. Δεύτερον, βία εναντίον των γυναικών. Αυτό έχει προκύψει ως ε, θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει το, έχει κάνει το πρόγραμμα Δάφνη με ανταλλαγή πολύ καλών ε, απόψεων και πολιτικών, αλλά οι πολιτικές ακόμη δεν έχουν ε, ενσωματωθεί, δεν έχουν εφαρμοστεί στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Πολλές φορές στα νέα κράτη-μέλη ζητήθηκε να υπάρξει η εκπόνηση τέτοιων πολιτικών. Υπάρχουν λοιπόν φιλοδοξίες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξουσιοδότηση να δράσει στους τομείς αυτούς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και ανισότητες στι αρμοδιότητες αυτές και ίσω είναι ώρα να επανεξετάσουμε το κατά πόσο υπάρχει επαρκή αρμοδιότητα έτσι ώστε να υπάρξει ένα νομικό εργαλείο για να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Σαφώ υπάρχει ανάγκη από την κοινωνία των πολιτών ω προ αυτό. Υπάρχουν φιλοδοξίε και προσδοκίε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. σω λοιπόν πρέπει να επαναξετάσουμε αν η στρατηγική τη Λισαβόνα ε, δίνει τη δυνατότητα για εκφώνηση κάποιε οδηγίε στον τομέα αυτό. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων. Πώς πρέπει να το πλαισιώσουμε τον ρόλο αυτό. Ο παραδοσιακό ε, ε, τομέας ε, της ισότητας είναι ένας που θα πρέπει να δράσουμε. Είναι σημαντικό, είναι παραδοσιακό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει και να αλλάξει. Είναι μια καλή βάση πολιτικής να πλησιωθεί δηλαδή στα πλέ, να γίνει όλο αυτό στα πλαίσια της ισότητας. Ένας πιο δυναμικός τομέας είναι η οικονομική ανάπτυξη. Εδώ Έχουμε δει πολλέ προσπάθειες για να υπάρξει mainstreaming σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων στα, θέματα της οικονομικής ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των γυναικών, ξέρουμε ότι χρειάζεται πλήρη συμμετοχή στις, ε, των γυναικών στην λήψη αποφάσεων και παρόλα αυτά στο αναθεωρημένα κείμενα για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική τα θέματα των δύο φύλων εξακολουθούν να είναι περιθωριοποιημένα. Ξέρουμε λοιπόν επί της αρχής τι συμβαίνει. Ίσως θα πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο πρακτικοί. Ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα αναδυόμενο πλαίσιο το οποίο αρχίζει να γίνεται όλο και πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και μελετούμε τα θέματα των, της ισότητας των δύο φύλων. Είναι ενδιαφέρον, είναι, γίνεται όλο και πιο σημαντικό για τους πολίτες και νομίζω ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι κίνδυνοι λόγω του τρόπου με τον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν θεσμοθετηθεί σωστά. Δεν έχουν θεσμοθετηθεί δηλαδή ως θέματα ίσης, ε, ε, διαχείρι... ίσης ε, μη διακριτικής μεταχείρισης και ισότητας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να θεωρήσουμε ότι όλα τα θέματα ισότητα των δύο φύλων μπορούν να εμπίπτουν στον γενικότερο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας μην ε, αφήσουμε λοιπόν τον παραδοσιακό τομέα της ισότητας. Έχουμε βέβαια και ε, ε, ίσως μικρότερου τομεί όπως ας πούμε η υγεία κτλ... αλλά πρέπει όλα αυτά να τα συνθέσουμε, να τα ενώσουμε, να τα συνδυάσουμε στα πλαίσια της ε, πρότασης που ίσως θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν. Το mainstreaming έχει αποτελέσει σταδιοίκη για την πρόθεση των θεμάτων ισότητας των δύο φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει πολύ προσεκτικά όταν λέει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και η εμπειρογνωμοσύνη αλλά και η εκπόνηση νέων πολιτικών για νέους τομείς. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε αυτό το διτό χαρακτήρα, γιατί πολλές φορές το ξεχνούμε και έχουμε μόνο τη διάχυση. Θα πρέπει να έχουμε και την κεντρική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά και την διάχυση όλων αυτών των αρχών σε διάφορους τομείς λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν διάφοροι τομείς στο mainstreaming που μπορούν να προχωρήσουν, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν προχωρήσει, ειδικά σε ό,τι αφορά την βία εναντίον των γυναικών, το gender budgeting επίσης, που είναι και αυτό τεχνική κομμάτι του mainstreaming. Υπάρχουν όμως και κάποια εξειδικευμένα θέματα. Θα υπάρξει κάποιο κονδύλι για τη νέα στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων. Θα είναι συγκεκριμένο δηλαδή κονδύλι που θα αποδίδεται στον τομέα αυτό έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και χρησιμοποιούνται μόνο για τον τομέα αυτό αντί να, είναι, να υπάρχουν γενικά κονδύλια που ίσως να μην εισρεύσουν στον τομέα αυτό. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε ποιος είναι, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το θέμα της ισότητας στο αποτέλεσμα. Να διευρύνουμε τους τομείς όπου, στους οποίους προχωράει η πολιτική αυτή, συμπεριλαμβάνοντας, για παράδειγμα, ε, επαρκή δεδομένα για την ε, βία εναντίον των γυναικών. Παρά, που, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, διάφορα σχέδια και προγράμματα για την βία εναντίον των γυναικών, δεν έχουμε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για να υποστηριχθούν οι σχετικοί δείκτες. Οπότε δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει την βία εναντίον των γυναικών ή αν οι πολιτικές αποτυγχάνουν ακόμη δεν έχουμε ούτε τις σχετικές αποδείξεις και πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα συλλογής δεδομένων για να ενισχυθούν αυτοί οι δείκτες. Ο δικός χάρτης περιλαμβάνει συγκεκριμένους τρόπους για να δούμε ποια είναι τα θέματα που εμπίπτουν στην ισότητα των δύο φύλων. Ο πιο σημαντικός ισχυρός τρόπος για να το δούμε αυτό είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο, ένα κατάλογος ο οποίος θα προωθεί τα θέματα αυτά, αντί να, τα, να βλέπει μεμονωμένα το κάθε θέμα. Ο δικός χάρτης ήταν εξαιρετική ε, κίνηση. Βασίστηκε στις υπάρχουσες πολιτικές ε, για την ισότητα των δύο φύλων ανά τον κόσμο, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. εγώ σας είπα πριν και για τα θέματα το, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η πολιτική ε, για, τη βία εναντίον των γενικών θα πρέπει να την λάβουμε πολύ πιο σοβαρά υπόψη μας, ένα πλαίσιο για την, για την ισότητα και πώς θα πρέπει αυτό να ενσωματωθεί στον γενικότερο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ καλύτερα από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Σίλβια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Τώρα θα ακούσουμε την καθηγήτρια Τζοβάνα Νταμολίν από το Πανεπιστήμιο του Μπάρι στην Ιταλία. Δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή να παρήστε μας σήμερα εδώ και να φέρω την εμπειρία μιας πανεπιστημιακής καθηγήτριας προς τους πολιτικούς. Έχω σκεφτεί πολύ το θέμα που συζητάμε προκειμένου επειδή η ειδικότητά μου είναι κοινωνική δημογραφία προσπάθησα να εντοπίσω ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στι οποίε πρέπει η Ένωση να αποδώσει την προσοχή. Φέτος είναι το ευρωπαϊκό έτος της καταπολέμησης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Φέτος λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη έκτακτε ανάγκε που έχουν σχέση με τον κίνδυνο φτώχεια και προβλήματα λόγω του φύλου. Ξέρουμε ότι οι γυναίκε είναι πιο εκτεθειμένες στη φτώχεια από ότι οι άντρε, ανάλογα με την ηλικία και την κοινωνική κατάσταση ιδιαίτερα. Θα ασχοληθώ λοιπόν ιδιαίτερα με τέσσερα σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι έκτακτη ανάγκη οι γυναίκες μόνες τους και ηλικιωμένες, οι γυναίκες που ζουν μόνες και είναι χωρισμένες, οι ντόνες που είναι μόνες μετανάστες και οι γυναίκες μόνες που υφίστανται βία στο σπίτι. Γυναίκες μόνες και ηλικιωμένες. Η γύρανση του πληθυσμού είναι σημάδι μιας βαθιάς δημογραφικής μεταβολής στις δυτικές χώρες άνευ προηγουμένου. Η ζωή όπως ξέρουμε επιμικίνεται και μάλιστα πολύ στις 19 από τις 27 χώρες της Ένωσης η, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες έχει ξεπεράσει τα 80 χρόνια. Η μακροζωία όμως δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για τη γυναίκα. Μερικές φορές οι γυναίκες που έχουν ξεπεράσει τα 65 χρόνια μένουν μόνες τους, είτε χωρισμένες, ε, είτε σε διάσταση, είτε χωρίς παιδιά, είτε χείρες και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις έχουμε φτώχεια και μεγάλη μοναξιά. Αυτές οι γυναίκες, φτωχές και ηλικιωμένε, στο μέλλον θα αυξηθούν σε αριθμό, στο βαθμό που αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Πώς μπορούμε τώρα εμείς να παρέμβουμε. Στόχος είναι σε νομοθετικό επίπεδο να φροντίσουμε όλες οι χώρες να δώσουν τη δυνατότητα στη γυναίκα να δουλεύει μέχρι τα 65 χρόνια με βάση τις ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες έτσι ώστε στο τέλος της ε, ζωής της εργασίας να έχουν μια πιο καλή σύνταξη γιατί πολλές φορές οι γυναίκες αυτές είναι σε συνθήκε φτώχεια. Με ειδικέ μελώτε που θα παρακολουθούν τι ανάγκε των ηλικιμένων γυναικών για κοινωνική υποστήριξη, υγειονομική υποστήριξη, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες που να βοηθάνε τις γυναίκες στο σπίτι γυναίκες που είναι μόνες και ηλικιωμένε, ιδιαίτερα αν έχουν και προβλήματα αναπηρίας γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν τέτοια προβλήματα στη μεγάλη ηλικία νέε μορφές επιχειρηματικής δράσης ε, υπέρ των ηλικιωμένων δηλαδή να βοηθιόνται τα πρόσωπα αυτά στο σπίτι τους δεύτερος στόχος αφορά τις γυναίκες που είναι μόνες και χωρισμένες γιατί έχουμε όλο και περισσότερα διαζύγια και ε, γυναίκες που ζουν χωρισμένες. Η αστάθεια αυτή στο γάμο οδήγησε σε αύξηση των αριθμών των μονογονικών οικογενειών. Γυναίκες δηλαδή με παιδιά. Στην Ιταλία, Φερρυπίν, μόνο τους εννοώ, στην Ιταλία στις δύο τελευταίες απογραφές είχαμε αύξηση 30% ανάμεσα στις δύο αυτές όσον αφορά τις μονογονικές οικογένειες με τη ρήξη των δεσμών του γάμου ε, επηρεάζεται το στυλ της ζωής και πολλές φορές η οικογένεια οδηγείται προς τη φτώχεια η μονογονική οικογένεια επιπλέον δε έχουμε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα στον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών που καθορίζεται και από τη φτώχεια και από το ότι πολλές φορές η μητέρα είναι απούσα γιατί δουλεύει προκειμένου να τα φέρει βόλτα. Βέβαια αυτό είναι μεταβατική φάση από τη στιγμή που η γυναίκα βρει ένα νέο σύντροφο ο οποίος θα αναλάβει και αυτός τις οικογενειακές ευθύνες με τον τρόπο του το βιωτικό επίπεδο επανέρχεται στο φυσιολογικό και το πρόβλημα φτώχειας για αυτού του είδους τις γυναίκες πάβει να υπάρχει. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες. Π.χ. Ε, δωρεάν νομική υποστήριξη στην περίπτωση που ο άλλος εταίρος ε, παραβιάζει τις συμφωνίες για τα παιδιά κλπ. Ε, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να επανέλθουν οι γυναίκες αυτές στην εργασία κυρίως για τις πιο νέες. Κίνητρα για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν γυναίκες μόνες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά. Μετά έχουμε τις μετανάστρες που ζουν μόνες τους. Η γυναικεία μετανάστευση σήμερα είναι μια πραγματικότητα που ακόμα δεν την γνωρίζουμε καλά. Γιατί είναι πολύπλοκη και έχει δύο μορφίες λόγω δύο προβλημάτων. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τη μετανάστευση κατά το φύλλο Μέχρι πριν από 10 χρόνια η μετανάστευση είναι φαινόμενο τυπικά ανδρικό. Οι, οι άντρες ψάχνανε δουλειά και από τη στιγμή που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα σχετικά σε μια χώρα η γυναίκα, η σύντροφό του, η μάνα των παιδιών ερχόταν και αυτοί μετά. Σήμερα το πλαίσιο αυτό έχει αλλάξει. Οι γυναίκε είναι πρωταγωνίστρες στη μετανάστευση. Είναι ένα νέο εταίρο, α το πούμε στο νέο πλαίσιο μετανάστευσης και η έκθεση του 2009 μας λέει ότι οι μετανάστες είναι το 49% της συνολικής μετανάστευσης στον κόσμο. Στην Ευρώπη το 52%. Και ευχαριστώ την προσοχή σας στις μετανάστες γυναίκες για τις 27 χώρες της Ένωσης που μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στο εσωτερικό της Ένωσης. Με βάση λοιπόν πρόσφατες στατιστικέ της Eurostat, πρώτες πρώτες είναι οι Πολωνίδε και οι Ρουμάνες. Αυτές είναι οι οποίε κινούνται με απόλυτη αυτονομία στο εσωτερικό της Ένωση. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι μετανάστριες συχνά βρίσκονται σε κατάσταση λεπτή, τρωτή, εκτίθενται στη φτώχεια περισσότερο από εκμετάλλευση στο χώρο εργασία κάνουν επισφαλή εργασία, χωρίς ε, συμβόλαια, χωρίς κοινωνική κάλυψη και υπόκειται φυσικά και στην κοινωνική περιθωριοποίηση και βία. Σε μερικές χώρες όπως η Ιταλία πρόσφατα μειώνεται, αυξάνεται πολύ ο αριθμός και ασχολούνται κυρίως με ως οικιακές βοηθοί, βοήθεια ηλικιωμένων, ε, ανάπηρων, άρρωστων, παιδιών. Η αύξηση της κινητικότητας που πολλές φορές από προσωρινή μετατρέπεται σε μόνιμη έχει επιπτώσεις στο δημογραφικό σκέλος όσον αφορά τις χώρες υποδοχής. Θα αλλάξει επίσης το πλαίσιο όσον αφορά τους γάμους γιατί έχουμε όλοι και πιο πολλούς μικτούς γάμους μεταξύ ντόπιου άντρε και ξένες γυναίκες. Ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες κοινωτικές χώρες και μεγάλη μία της γονιμότητας που μειώνεται μεν στις χώρες προέλευσης αλλά αυξάνει στις χώρες υποδοχής. Αυτό είναι ένα νέο δημογραφικό στοιχείο. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά. Να ξεπεραστεί η διπλή άνηση μεταχείριση τις οποίες ε, θύματα είναι οι γυναίκες μετανάστριες ώστε να τον κίνδυνο φτώχεια και του φύλου. Να ξεπεραστεί το εμπόδιο της επικοινωνίας με το να μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας παραμονής με ειδικά μαθήματα και να υπάρχει και ο γλωσσικός και διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Να έχουμε συγκεκριμένα μαθήματα κατάρτισης, ειδικά για τις ξένες γυναίκες, ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, παραδείγματο χάρη στην Ιταλία, νοσικόμες, γυναίκες οι οποίες βοηθάνε τα παιδιά, να υπάρχουν ειδικά μαθήματα για αυτές. Κάλυψη για δουλειά, να υπάρχει μια ειδική κάρτα υπηρεσιών, να υπάρχουν δυνατότητες ε, να προσφύγουν οι γυναίκες αυτές αν έχουν μια άμεση ανάγκη και να δοθεί προτεραιότητα σε προγράμματα ενσωμάτωσης των μεταναστριών. Πέρα από τα συγκεκριμένα προγράμματα υπέρ των μεταναστριών πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κίνηση εποπτείας του φαινόμενου κινητικότητας. Δεν έχουμε στοιχεία. Χρειαζόμαστε και επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη γυναικεία μετανάστευση με τράπεζες δεδομένων κατά εθνικότητα κατά με τη δυνατότητα εργασίας, αμοιβή των γυναικών και δείκτες, όπως είπε η Αγγλίδα συνάδελφος, δείκτες φτώχειας και κυρίως να ακούμε τις ενδιαφερόμενες με ερωτηματολόγια. Και ένα τελευταίο σημείο, αν έχω λίγο χρόνο, είναι γυναίκες που ζουν μόνες τους αλλά εφίστανται βία στο σπίτι όπου ζουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Εκ μέρους του συζύγου ή εκ μέρους ενός άλλου μέλους της οικογένειας προερχόμενη η βία. Είναι δύσκολο η βία που υπόκειται η βία να αφήσει το σύντροφό τη. Είναι παράδοξο, αλλά γυναίκα εξακολουθεί να αφησει το συντροφο τη ειναι παραδοξο αλλα η γυναικα σου να αγαπαει τον άντρα ακόμα και όταν υφίσταται βία. Και πολλέ φορέ υφίσταται πίεση να μείνει στην οικογένεια και από τον σύντροφό της αλλά όταν η βία είναι σαφής και από τους άλλους τα άλλα μέγη της οικογένειας επ' αυτού μερικές ιδέες και τελειώνω ε, αν θέλετε σταματάω εδώ τα έχω γράψει στο κείμενό μου μπορείτε να διαβάσετε ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Νταμολίν. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Μαρίσα Σολέτο, που είναι διευθύντρια του Ιδρύματος για τις Γυναίκες ε, στην Ισπανία. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως ε, που ήρθα σήμερα να σας μιλήσω. Είμαι διευθύντρια μιας μη κυβερνητική οργάνωσης που έχει ως ε, απότερο στόχο τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές για την πρόθεση των πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια καθώς και με τις διάφορες αυτόνομες περιοχές ε, για να εκπονήσουμε προτάσεις και νέα εργαλεία για την προώθηση της ισότητας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες που προέρχονται από τις γνώσεις που έχουμε για την κατάσταση και από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε στο Ίδρυμά μας. Ξέρετε τελικά η παρέμβαση που είχα προετοιμάσει ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις ε, παρουσιάσεις των συναδέλφων. Έχουμε τον οδικό χάρτη και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των δύο φύλων ε, που ισχύουν και υπάρχουν κάποια έγγραφα αξιολόγησης ε, από πλευράς της Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου. Και τι προκύπτει ότι παρά την πρόοδο που ε, έχουμε σημειώσει σε αυτό το τομέα, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Απασχόληση, συμμετοχή στα κοινά, οικογενειακά βάρη κτλ. Οι προτεραιότητες και οι στόχοι δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. Τα προβλήματα που είχαμε παραμένουν δυστυχώς ακέραια. Το σημαντικότερο είναι να θέσουμε σαφέστατους στόχους όταν προετοιμάζουμε νέες στρατηγικές. Αν θέλουμε ε, μεσομακροπρόθεσμα να είναι λυσίτελης, Ο στόχος του προγράμματος εργασίας 2006 έως 2010 εστιάζει στην ε, συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή, στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ε, την ε, κατάργηση της βίας κατά των γυναικών, την κατάργηση των στερεοτύπων, πολιτική ισότητας, αναπτυξιακή πολιτική, Όλα αυτά είναι απαραίτητες συνιστώσεις ε, μιας νέας στρατηγικής. Θα ήθελα να σχολιάσω περαιτέρω ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία που αντιστέκονται στις αλλαγές, παραμένουν αναλύωτα. Παραδείγματος χάρη, Α πάρουμε τις γυναίκες μέσα στον ιστό των επιχειρήσεων. Τι εννοώ, ε, δυνατότητα επιχειρη ε, εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και δυνατότητα ε, κατάληψης υψηλών θέσεων μέσα στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένας κοινωνικός δείκτης και δυστυχώς δεν σημειώνεται μεγάλη πρόοδος. Βεβαίως έχουμε την οικονομική κρίση αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε να υποβάλουμε προτάσεις ε, όπως και τα τελευταία χρόνια για να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις ε, ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες ε, στο χώρο εργασίας. Δεν θα τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας εάν δεν προτείνουμε διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ε, επιχειρήσεων και των θεσμικών οργάνων. στο επίπεδο των επιχειρήσεων αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός γυναικών και κυρίως τις υψηλές θέσεις. Και ξέρετε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια ευκαιρία που πρέπει να δράξουμε η οικονομική κρίση. Ξαναλέω ότι μας αφορά η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα στις ανώτερες βαθμίδες των επιχειρήσεων. Δεν είναι βέβαια νέα αυτή η πρόταση, πρέπει όμως να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών στην καθημερινή ζωή, διότι παραμένουν αντιμέτωπε ε, με πολλές δυσκολίες οι γυναίκες, η κατάσταση είναι σοβαρή και χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική κυρίως ε, για την βία που πλήττει τις γυναίκες. Οφείλουμε να ερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο με καλύτερο τρόπο. Δεν ξέρουμε καν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φαινομένου αυτού στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να έχουμε ομοιόμορφα εργαλεία, ομοιόμορφους ε, ορισμένε αποφάσεις. Εάν γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο βάθος το φαινόμενο, τότε θα μπορέσουμε να προτείνουμε στρατηγικές ε, που θα προστατεύουν καλύτερα τα θύματα. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε προληπτικές ε, δράσεις αποτελεσματικές. Ε, η ιδέα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την εκπόνηση δικτών που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλή. Επίσης προτείνονται μέτρα διασυνοριακά, διακρατικά για την προστασία των θυμάτων. Επίσης ε, εντάλματα για την προστασία των θυμάτων πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι όπως καταλαβαίνετε σημαντικό να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών και πάλι εδώ τίθεται αυτό το ε, ακαθόδε ζήτημα της άδεια μητρότητας και της άδεια πατρότητας. Χρειάζεται ισότιμη κατανομή των ευθυνών μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Εδώ και δεκαετίες ζητάμε από τους άντρες μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών. Ωραία. Ας περάσουμε από τα αιτήματά μας σε κάποια νομοθετική δράση. Οι κανόνες ε, που επιτρέπουν τη χορήγηση άδεια ε, μητρότητα και πατρότητας ε, πρέπει να διακρίνονται από σαφήνεια και να καταργήσουμε η αδίποτε κοινωνική διαφοροποίηση ως προς την χορήγηση αυτών των αδειών ε, μητρότητας και πατρότητας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να προβλέψουμε ένα χρονοδιάγραμμα που θα κατοχυρώνει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο είδη αδειών. Κατόπιν, η μέθοδοι ενσωμάτωσης στα κράτη-μέλη, ε, η οριζόντια προσέγγιση της πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων, δηλαδή πιστεύω, ότι χρειαζόμαστε δημιουργία εργαλείων ούτω ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Η ισότητα των φύλων πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι ε, πολιτικές σε κρατικό επίπεδο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή τη διάσταση και στα θεσμικά όργανα τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση διότι ε, είναι θέμα κοινωνική ποιότητα. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και μέσα στο κοινοτικό και εκτιμένο. Το ζητούμε εδώ και χρόνια. επίση είναι ένα δείκτη σχετικά με την ε, λειτουργία του ευρωπαϊκού Συστήματο. Ε, είναι ένα πάγιο αίτημά μα. Ε, παρόλα αυτά, πρόοδο δεν έχει σημειωθεί ούτε στα κρατημέλη, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον εγώ αυτό πρεσβεύω. Ε, νομίζω ότι είναι θέμα συντονισμού σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα κράτη-μέλη νομίζω ότι οφείλουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω αυτό το θέμα και να προτείνουμε συγκεκριμένες μεθόδους ενσωμάτωσης ε, της διάσταση της ισότητας των δύο φύλων στις πολιτικές ε, και να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα ώστε να επιτύχουμε την ομοιομορφία των επιμέρους πολιτικών. Το budgeting, η, ε, η λήψη υπόψη της διάστασης των γυναικών στον προϋπολογισμό κάθε εξεχωριστής πολιτικής, κάθε δραστηριότητας εθνικής και ευρωπαϊκής είναι κάτι το απαραίτητο. Τα φορολογικά συστήματα οφείλουμε να τα αναθεωρήσουμε επίσης, ούτως ώστε να μελετήσουμε διεξοδικά ποια μέτρα φορολογικά αποτελούν την ε, είσοδο ε, των ε, γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι πολιτικές απασχόλησης, ναι, μεν επιμένουν στη συμμετοχή των γυναικών, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν οικονομικές πολιτικές που ανερουν τις πολιτικές απασχόλησης. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια. Οφείλουμε να καταργήσουμε αυτές τις ανακολουθίες. Ξαναλέω επίσης ότι είναι θέμα κοινοτικού και Πρέπει να ενσωματώσουμε αυτή την διάσταση στο κοινοτικό και εκτιμένο ε, και στην νομοθεσία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία των οργάνων της Ένωσης και πρέπει να επιμένουμε ούτω ώστε να διατηρηθούν οι προτεραιότητες που έχουμε ήδη ορίσει. Ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρο, Θα ακούσουμε άλλες τρει ε, παρεμβάσεις και μετά θα κάνουμε μια κάπως γενικότερη συζήτηση. Να ευχαριστήσω τις ε, ομιλήτριές μας. Θα τις ξανακούσουμε εξάλλου γιατί θα τεθούν ερωτήσεις από τους παρισταμένους. Η αντιπρόεδρος μας θα πάρει πρώτη το λόγο, η κυρία Γιαρόκα. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, ε, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. I'm going... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Και θα είναι εύκολο αυτό, γιατί πολλά από όσα ήθελα να πω ακούστηκαν ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική εισαγωγή. Είναι χαρά μου που είμαι η σκιώδη γιατί πέρα από τα γενικά θέματα τα οποία συζητούμε και τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί πολύ σωστά, φαίνεται και από τη δουλειά της Επιτροπής ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά τώρα έχουμε και την ε, δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα έξι σημεία του οδικού χάρτη και στην Επιτροπή αλλά και βλέπω ότι και οι ευρωγνώμονε ε, καταδεικνύουν κάποιου νέους ε, τομεί ε, που αναπτύσσονται και που εμπλουτίζουν τη συζήτησή μα και την εμβαθύνουν. Για τα όσα υπόθηκαν, θα ήθελα σύντομα να σχολιάσω και να αναφέρω και κάποια νέα στοιχεία ως σκιώδης συγκήτρια της έκθεσης ως πρόβλημα εγώ αναγνωρίζω και την χαμηλή εφαρμογή των ε, υπαρχουσών ε, οδηγιών. Αυτό φαίνεται στις ανατολικές κυρίως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρηκα πολύ που ακούστηκε το θέμα από την ε, κυρία Γουόλμπι, γιατί δεν έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ως, προς, ως, προς, ως τώρα για την για, τις κοινωνικές, για τους κοινωνικές Ο Επίτροπο Σπίτλε είχε ε, εισαγάγει το νέο δικό χαρτί και ήταν πολύ ικανοποιητικό το γεγονό ότι είχαμε έτσι ένα υποθέμα γιατί θεωρούσαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο με το πρόβλημα θα έριχνε φως σε τομεακά προβλήματα όπως ας πούμε ε, το, της, τη διακριτική μεταχείριση της οποίας την χάνουν οι γυναίκες στην Ευρώπη. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν ήταν θεματικά στον τομέα αυτό αλλά τουλάχιστον ε, ξεκινήσαμε να κατανοούμε τι ακριβώς σημαίνει η διακριτική μεταχείριση και τονίσαμε την ε, διακριτική μεταχείριση σε διάφορους τομείς γιατί οι γυναίκε πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ, διαφορετικά, πολύ διαφορετική διακριτική μεταχείριση από του άντρε. Αναγνωρίζοντα λοιπόν αυτή τη ε, διαφορά και βάζοντα και αυτό τον παράγοντα στην εξίσωση, τώρα ήρθε η ώρα να καθορίσουμε την πολιτική σύμφωνα με το gender mainstreaming ώστε να αντιμετωπίσουμε τη διακριτική μεταχείριση που, οποία οποίας χάνουν οι γυναίκες. Σημαντικό επίσης για μένα είναι να κάνουμε τους πολίτες να κατανοήσουν ότι ε, επενδύοντας άμεσα στις ε, ε, οικονομικές, στους οικονομικούς τομείς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να μειωθούν οι ανισότητες. Βέβαια πολλοί θεωρούσαν ότι θα γίνει το αντίθετο, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Οι γυναίκες δεν έχουν ε, μεγάλη πρόσβαση στην εκπαίδευση πάντα ή στον τομέα της υγείας. Και είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε αυτό στα πλαίσια του έτους για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής. Έχουμε τα νέα στατιστικά από τη Eurostat για το πώς αναπτύσσεται, όσο αυξάνεται η ε, φτώχεια στην Ευρώπη. Εγώ έχω μελετήσει και τους δείκτες και δείχνουν πραγματικά σαφέστερα το πώς έχει η κατάσταση. «16% Τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πλήττεται άμεσα από τη φτώχεια, από την ένδια. Εγώ στη δική μου χώρα όμω, πρέπει να σα πω ότι ένα τρίτο του των πολιτών ζουν ε, κάτω από τα, από τα όρια της φτώχειας, ένα τρίτο είναι εθνικές μειονότητε, που σημαίνει δύο τρίτα του πληθυσμού μας βρίσκεται σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Είναι πραγματικά αυτοί που πλήττονται περισσότερο και την χάνουν και των μεγαλύτερων διακριτικών, της μεγαλύτερης διακριτικής μεταχείρισης. όπως είπε και η κυρία Νταμολίν, υπάρχουν και, άλλοι, και άλλες ομάδες γυναικών που πλήττονται σημαντικά. Όχι μόνο ηλικιωμένε, όχι μόνο αυτές που ε, είναι γονείς, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που έρχονται από βγαίνουν από ορφανοτροφία και δεν έχουν βρει έναν τρόπο να ζήσουν μέσα στην κοινωνία. στο παιδικό σταθμό του παιδιού μου, κάποια παιδάκια, ένα παιδάκι, ένα αγοράκι δύο χρονών, το πήγαν στο ορφανοτροφείο και ρώτησα γιατί και γνώρισα τη μητέρα και ήταν ένα κορίτσι 22 χρονών. Είναι μόνη μητέρα, έχει μικρό παιδί, είναι ανεργή, είναι, ανήκει στο Ρώμα, ε, έρχεται από ορφανοτροφείο, δεν έχει ε, οικογένεια, 22 χρονών, είναι άστεγη και έχασε το παιδί της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά στέλνονται σε ορφανοτροφία σε αυτή την πολύ ευτυχισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι γυναίκες αυτές δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το νοδικό χάρτη να ενισχυθεί αυτή η διάσταση. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιαρόκα. Η κυρία Κορνέλισεν τώρα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλες τις ε, προσκεκλημένες ε, ειδικού στο θέμα. Θα αναφερθώ σε μερικά σημεία που τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή μας όσον αφορά τη νέα στρατηγική. Άκουσα με πολύ περιεργία τη φράση ότι η στρατηγική της Ένωσης είναι πιο καλή στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απέσια η κατάσταση στα άλλα μέρη του κόσμου. Η στρατηγική για τα φύλλα στην Ευρώπη πάσχει από ωραία λόγια και έλλειψη συγκεκριμένων πράξεων. Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι στην πράξη, η πολιτική για την ισότητα, ναι μεν λέμε ε, ότι πρέπει να μπει το στοιχείο αυτό στις εξωτερικές δράσεις της κοινότητας. χάρη βλέπουμε τι έγινε με το σεισμό στην Αϊτή. Πολύ βοήθεια στάλει προς τη χώρα αυτή. Αλλά βλέπετε στην τηλεόραση άντρες βλέπουμε να δίνουν μάχη γιατί η λίγη ποσότητα νερού και τροφίμων και οι γυναίκες είναι στο περιθώριο, πίσω τις βλέπουμε. Ακούμε για πάρα, πολλούς, πάρα πολλά θύματα βιασμών. Στην όλα αυτά σήμερα. Και οι γυναίκες ε, μάχονται μεταξύ τους εναντίον μιας της άλλης για το λίγο νερό. Αυτό η Ένωση που έστειλε τη βοήθεια εκεί δεν το αντιμετώπισε ως πρόβλημα. Στην πράξη όλα αυτά. Στην πράξη πάσχουμε λοιπόν. Άλλο παράδειγμα, χθες διαπίστωσα ότι έχουμε, γίνεται μια συζήτηση για την άδεια λογομητρότητας. Θα ψηφίσουμε κάτι τέτοιο στην Επιτροπή Απασχόλησης στο Κοινοβούλιο. Όλοι μεν είμαστε υπέρ να μην υφιστάνει σε μεταχείριση στην αγορά εργασία σε βάρο των γυναικών, αλλά όταν φτάσει ο κόμπο στο χτένι, τελικά τα συμφέροντα της επιχείρησης πρωτεύουν και διαγράφει μία παράγραφος που αντιστρέφει το βάρος τη απόδειξης. Όταν δηλαδή ένα ε, επιχειρηματίας θέλει να απολύσει μία γυναίκα που είναι έγκυα. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρακτικά μέτρα οι γυναίκες και η κρίση. Πολύ σημαντικό θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον πληθυσμό ο οποίος γυράσκει. Άτομα που θα χάσουν τη δουλειά τους σήμερα, που δεν θα είναι στην αγορά εργασίας στο μέλλον, πώς θα το ισοφαρίσουμε αυτό, πώς θα βρούμε δηλαδή έναν τρόπο από τη μια μεριά το πώς θα μοιάζει η κοινωνία και η αγορά εργασίας 20 χρόνια από σήμερα και πώς θα προετοιμαστούμε με μέτρα να είμαστε έτοιμοι για αυτό το φαινόμενο. Φορολογική στρατηγική, πολύ σημαντικό θέμα. Στην Ολλανδία για πολλά χρόνια είχαμε φορολογικές ρυθμίσεις που ενθάρρυναν τις γυναίκες να μείνουν στο σπίτι, να φροντίζουν τα παιδιά. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Και μια τελική παρατήρηση. Πολλά, πολλά σημεία τα παραλείπω γιατί δεν έχω χρόνο. Ανάγκη για έρευνα, για τη βία και για κάθε άλλη μορφή που σχετίζεται με τα φαινόμενα αυτά. Σε μερικές χώρες οι γονείς φροντίζουν πολύ περισσότερα τα παιδιά από τις άλλες χώρες. Γιατί, ποιες είναι οι παράμετροι για αυτό το φαινόμενο. Χρειαζόμαστε δείκτες και παραμέτρους. Στην Ολλανδία πληρούνται όλα τα κριτήρια της Λισαβόνας για την απασχόληση των γυναικών. Αλλά τελικά δεν έχει σημασία να δουλεύουν 2 ή 12 ώρες τη εβδομάδα. Η απασχόληση των γυναικών στην Ολλανδία δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική ανεξαρτησία. Πρέπει τα νούμερα να τα βάλουμε στη σωστή προοπτική και να έχουμε τους σωστούς ορισμούς. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα όσα μας είπατε και θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία αυτά για την έκθεσή μας. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κυρία Κορνέλισεν. Η κυρία Μπελίντα Πάικ θα πάρει το λόγο τώρα, διευθύντρια αρμόδια μεταξύ άλλων για τα θέματα ισότητας από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόλησης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση και ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις που καταθέτουν ε, οι παρισταμένοι. Και πέρα από το τι συμβεί σήμερα στην Επιτροπή θα έχουμε και τις εργασίες της Ολομέλειας. Θα ήθελα να πω κάτι για το γενικό πλαίσιο. Πρώτον, αναφέρθηκαν οι ομιλήτριε σε ελαφρύ αλλαγέ που έχουν γίνει στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πώ χειριζόμαστε τα θέματα ισότητα. Πέρα από τις αλλαγές υπάρχει μεγάλη συνέχεια. Θα ήθελα να σας το εξηγήσω. Η δικιά μου υπηρεσία ασχολείται με την κατάρριξη της διακριτικής μεταχείρισης και την πολιτική της ισότητας και ανήκουμε στην Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και η Επίτροπός μας θα είναι αυτή που θα είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ηθαγένεια, για την ισότητα. Ε, αυτό μας επιτρέπει να έχουμε στενή σχέση με την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Τα θέματα ισότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά να ενταχθούν σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά έχουμε το προβάδισμα γιατί είμαστε στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τις κοινωνικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων χειριζόμαστε και το ΕΚΤ. Τώρα ε, με το νέο χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολούμαστε και με άλλες πτυχές κοινωνικής πολιτικής ε, και έχουμε ισχυρή επικοινωνιακή πολιτική ε, και συνεργασία με τους συναδέλφους από τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ε, όλοι τόνισαν πόσο βασική προτεραιότητα είναι η διεπηρεσιακή συνεργασία. Η Επίτροπος μας ε, ασχολείται ε, γενικότερα με τα θέματα ισότητας και πιο συγκεκριμένα με τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών. Προς το παρόν, όπως ξέρετε, υπάρχουν συμπεράσματα που συζητώνται στο Συμβούλιο για την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών που πρότεινε η Ισπανική Προεδρία. Στις 8 Μαρτίου αναμένεται η έγκρισή τους. Είμαστε στην συνεργασία με τους συναδέλφου Δικαιοσύνη εσωτερικών υποθέσεων. Η νέα Επίτροπο έχει αναλάβει ισχυρότατη δέσμευση σε αυτό το τομέα. Άρα θα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες από τη νέα δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο βαθμό που θα επιλέξετε εσεί να ορίσετε τη νέα Επίτροπο. Έτσι είναι το δικαίωμά σα, το θεσμικό σα δικαίωμα. Ε, θα ήθελα να ακούσουμε παρεμβάσεις και ερωτήσεις από όλους, οπότε θα είμαι σύντομη για το, την παρακολούθηση ή τη συνέχεια του οδικού χάρτη. Με το νέο πρόγραμμα του κυρίου Μπαρόζο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ε, υποθέτουμε ότι θα υπάρξει μια συνέχεια με τη στρατηγική όπως το ονομάσουμε, όπως ονομάσουμε τη νέα πολιτική στρατηγική μάλλον θα λέγεται. Πέρυσι στο Στρασβούργο έγινε διευρυμένη συνεδρίαση ε, όλων των επιτροπών που ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα για να δούμε πώς ακριβώς έχει υλοποιηθεί ο εφιστάμενος οδικός Χάρτη και να εντοπίσουμε τις προτεραιότητες για τις μελλοντικές δράσεις ενός μελλοντικού οδικού χάρτη. Κυρίως ε, στα πλαίσια της οικονομικής ε, κρίσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς τι έχει αλλάξει από την ε, από τη στιγμή που εκπονήσαμε την περασμένη στρατηγική. Ε, αναπόφευκτα ε, ή μάλλον ε, τι να πω, δυστυχώ ε, οι ίδιε παραμένουν οι προτεραιότητε. Υπάρχουν και κάποια νέα στοιχεία, αλλά πάντοτε χρήσιμο είναι να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στι συγκυρίε οικονομικέ ή τι κοινωνικέ. Αυτό είναι το εφαλτήριό μα. Κατόπιν, κάναμε μια διευρυμένη διάσκεψη με του κοινωνικού εταίρου και όλου του ενδιαφερόμενου φορεί πέρσι και συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις και η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα των Δύο Φύλων όπου συμμετέχουν οι εθνικοί αρμόδιοι φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι, συνέχισαν τις εργασίες ε, και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το έργο τους και όλο αυτό το υλικό ε, να το διαβιβάσουμε στην εισηγήτρια και στην Επιτροπή για να σας επικουρήσουμε κι εμείς. Τώρα, άλλο σημαντικό υπόβαθρος προς τις εργασίες μας ε, ε, μόλις ε, μας μοιράστηκε η περίληψη του σχεδίου δράση για την υλοποίηση της πλατφόρμας του Πεκίνου. Η Σουηδική Προεδρία, να σας υπενθυμίσω, τους τελευταίους μήνες ε, συνέταξε μεγάλη έκθεση για την πλατφόρμα Πεκίνου ΣΥΝ 15 εξετάζει τις δραστηριότητες σε κάθε τομέα, οπότε είναι πάρα πολύ καλή και περιεκτική έκθεση. Σας συνιστώ να τη διαβάσετε. Ε, τον Ιούλιο σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τη νέα στρατηγική μας και είναι πάρα πολύ καλό που θα έχετε ολοκληρώσει την έκθεσή σας τον Μάιο και δεν θέλουμε να υπερβούμε τον ε, Ιούλιο γιατί ξέρουμε ότι ε, η Βελγική Προεδρία θέλει να επεξεργαστεί την πολιτική και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να, για να αναλυφθούν συγκεκριμένες δράσεις. Πάντως θα βασιστούμε στη δράση και στην πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα μεριμνήσουμε ώστε να έχει μια εξωτερική διάσταση η νέα ε, στρατηγική. Δηλαδή να μην υπάρχουν ανακολουθίε ε, στα μηνύματα που περνάμε στου εταίρου μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό, σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε. Επίση, ε, υπάρχουν και το θέμα τη διακυβέρνηση. Ποιο κάνει τι. Και λοιπόν ε, αυτό μας ε, οδηγεί στη δράση των θεσμικών οργάνων. Είπαμε, ανέλαβε δέσμευση η Βελγική Προεδρία ήδη ε, να εγκρίνει συμπεράσματα για τη νέα στρατηγική και ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει στη δυνατότητα για την Ουγγρική Προεδρία, το, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ένα δωδεκάμινο, να αποφασίσει ναι, ενίσχυση της Συμφωνίας Συμβουλίου για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Γιατί ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ στην Επιτροπή σας. Ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ε, πρέπει να συσπηρωθούν όλοι, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υφιστάμενες δομές και όλα τα υφιστάμενα μέσα. Ε, και να έχουμε υπόψη το τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην χάσουμε καμία ευκαιρία να εντάξουμε σε άλλους στόχους στρατηγικών το θέμα της όντας των δύο φύλων. Η ανάκαμψη για το 2020 ε, τη, κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας τονίστηκε πως η ισότητα των δύο φύλων συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και το ίδιο μας είπε ε, και συνάδελφος Γιαρόκα. Ε, πρέπει και εμεί ε, να μεριμνήσουμε ώστε να συνεχιστούν οι συζητήσει για τη συμμετοχή τη ισότητα των δύο φύλων στο σχέδιο 2020. Υπάρχει και το σχέδιο δράση τη Στοκχόλμη που πρέπει να μα απασχολήσει και άλλοι τομεί για την ένταξη των Ρώμα, για την, ε, τα άτομα με αναπηρίες, δημογραφική γύρανση, που θα προκύψουν από το νέο σχετικό πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ώστε να ενταχθεί το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων σε όλες αυτές τις στρατηγικές. Η νέα στρατηγική πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα για τα επόμενα πέντε χρόνια βάσει του οποίου θα, στους τομείς κλειδιά ε, θα εντάξουμε σε όλους τους τομείς λοιπόν το ζήτημα των δύο ε, Και τα βασικά ζητήματα τι είναι οι διαφορές τους ε, μισθούς και υπάρχει μεγάλη μορφή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα στους μισθούς. Δεύτερον, βία κατά των γυναικών είναι Βέβαια όλα φαίνονται απλά, έτσι λέμε δύο τίτλους, αλλά ξέρετε πώς να γίνουν οι μετρήσεις, ε, πώς να διαπιστώσουμε ακριβώς ποιος κάνει τι, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτές είναι οι κατάφορες πάντως ανισότητες ε, που διαπιστώνουμε μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ισότητα των δύο φίλων και πώς επηρεάζει αυτό τους άντρες στην συμφιλίωση οικογενειακής και της επαγγελματική ζωής τονίσαμε ότι οι άντρες για διάφορους λόγους δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που έχουν για να συμφιλιώσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή τους. Δηλαδή δεν ζητάνε άδεια τόσο όσο οι γυναίκες. Ε, γι' αυτό είναι καλό να έχουμε αυτή τη νέα οδηγία ε, που προέκυψε από τη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων. Ε, και γιατί αυτό σημειώνεται σε κάποιους επαγγελματικούς κλάδους. Εφόσον λέγαμε πώς να κατέχουν υψηλά αξιώματα οι γυναίκες, να ασχοληθούμε και με το πω γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άντρες δάσκαλοι, ας πούμε, και το αντίθετο. Ε, στις επόμενες ε, γενιές ε, θα πρέπει τα παιδιά να βλέπουν και οι επόμενες γενιές να βλέπουν ότι ναι οι γυναίκες έχουν υψηλά αξιώματα σε επιχειρήσεις αλλά και οι άντρες είναι δάσκαλοι. Ευχαριστούμε κυρία Πάικ. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν ερωτήσεις και να σχολιάσουν τα θέματα που μας απασχολούν παρακαλώ να είναι σύντομες οι ερωτήσεις σας. Μην κάνετε δηλώσεις, υποβάλλετε σύντομες ερωτήσεις, ούτως ώστε τα μέλη της ομάδας να έχουν ε, την δυνατότητα να απαντήσουν. Η κυρία Γκαρσία Πέρες θα πάρει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τις προσκεκλημένες μας που μας μίλησαν με τόσο ενδιαφέροντα λόγια. Έχουμε μπροστά μας μία πραγματικότητα με την οποία όλοι συμφωνούμε. σχετικά με την κατάσταση για την ισότητα ανδρών γυναικών. Μερικές φορές μπορεί αυτό να μας δημιουργεί απογοήτευση. Δηλαδή μιλάμε συνέχεια ποια είναι τα από τα εμπόδια, τα κολλήματα, τι προβλήματα συναντά η ισότητα ανδρών και γυναικών. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε πρώτον τι πετύχαμε στο παρελθόν προκειμένου να συνεχίσουμε το δρόμο της ισότητας ανδρών και γυναικών με πρόοδο. Και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και τις προσπάθειές μας στα εργαλεία ελέγχου που επιτρέπουν την υλοποίηση της ισότητας ανδρών Έχουμε νομοθεσία, έχουμε εργαλεία. Ας δούμε πώς θα κινήσουμε και άλλους μηχανισμούς ελέγχου για το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά, όπως η καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων. Έχουμε εμπειρίε από τις χώρες μας σχετικά. Τώρα για τις εξηγήσεις που μας έδωσε και η κυρία Μπερίντα Πάικ σχετικά με τις αρμοδιότητες σε θέματα ισότητας και πώς γίνεται η κατανομή τους στην Κομισιόν. Έχω μία ερώτηση προς τις εισηγήτριές μας. Θεωρείται αναγκαίο η Κομισιόν παραδείγματο χάρη, αλλά θα μπορούσαμε να κατέβουμε το σε επίπεδο και να πάμε στις χώρες μέλη, σε άλλου είδους όργανα και θεσμούς. Να υπάρχει ένας μόνος οργανισμός που να προωθεί, να συντονίζει, να εποπτεύει τα θέματα αυτά όλων των επιμέρους πολιτικών για την ισότητα διότι είναι σημαντικό το εγκάρσιο στοιχείο αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δημόσιο όργανο κατά να εποπτεύει την εφαρμογή όλων αυτών των πολιτικών για την ισότητα. Πρόεδρος, Η κυρία Παπάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Κομισιόν για τη δημογραφική κρίση. Ένα παράδειγμα. Για το 2010 στη Βουλγαρία έχουμε 65% ε, συνταξιούχων γυναίκες και 35% άνδρες στη σύνταξη. Μεταξύ των κρατών μελών έχουμε 10 χρόνια διαφορά στο προσδόκιμο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και το 2030 θα έχουμε επιπλέον 30 εκατομμύρια συνταξιούχους στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό, ότι η δημογραφική κρίση είναι ένα σημαντικό θέμα φίλων. Και όπως ακούσαμε, είναι πολύ αρνητικό να είναι κανείς γυναίκα και ηλικιωμένη στην Ευρώπη. Και ρωτώ, η Κομισιόν θα αναθεωρήσει τον οδικό χάρτη με βάση αυτή τη δημογραφική εξέλιξη, ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέματα αύξησης τη ηλικία του φύλου για πρόσβαση στι ιατρικές υπηρεσίες, στις κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες αυτές που ήδη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Προέδρο. η κυρία Τόμψεν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις ομιλήτριες όλα όσα μας είπε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η κυρία Βάλπη αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε η κυρία Βάλπη ότι ως γυναίκες εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, δεν επηρεάζουμε το επίπεδο αυτό. Πρέπει να βελτιωθεί ο ρόλος των γυναικών σε αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στα ανθρώπινα δικαιώματα. σε σχέση με την ισότητα των φίλων και το mainstreaming. Γιατί τι βλέπουμε στην Ευρώπη. Το 2002 η Ένωση ε, ενέκρινε μια οδηγία για θέματα φίλου, όπου έλεγε ότι κάθε χώρα θα πρέπει να έχει ένα Ινστιτούτο για το θέμα των φύλων. Ευρωπαϊκό όργανο έχουμε, αλλά στις χώρες μέλη δεν έχουμε πια ένα τέτοιο Ινστιτούτο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το Ινστιτούτο αυτό συγχωνεύτηκε με άλλες 7 7-8 Ινστιτούτα που υπήρχαν και δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα των φίλων λοιπόν πέρασε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μόνη χώρα στην Ευρώπη που ακόμα έχει Ινστιτούτο De la Mujer για τη γυναίκα είναι η Ισπανία στις άλλες χώρες έγινε αυτή η συγχώνευση όπως σας είπα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πλεονέκτημα για τις γυναίκες να ενταχθεί το θέμα του στα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί φυσικά εκεί υπάρχουν περισσότερα κονδύλια Αλλά όπως είπε η κυρία ε, Γιαρόκα για τις γυναίκες Ρώμα υποφέρουν από άλλου είδους καταπίεση από ότι οι άνδρες Ρώμα. Το ίδιο πράγμα για τα άτομα που έχουν ε, προβλήματα αναπηρίας κλπ. Ή ανήκουν σε μια μειονότητα και είναι γυναίκες. Θα ήθελα μερικά επιπλέον σχόλια πάνω σε αυτό αν γίνεται. Τέλος για την ε, καθηγήτρια ε, Δεμολίν. Πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε με αυτές τις ε, τροτές, ας το πούμε, ομάδες γυναικών στη χώρα μας. Γιατί οι γυναίκες ζουν όλο και περισσότερο. Η ομάδα αυτή γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Μεταξύ των ηλικιωμένων η ομάδα των γυναικών εννοώ. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε για γυναίκες που ζουν μόνες τους ή που είναι ε, χωρισμένες. Αν βρουν έναν νέο εταίρο, ε, σύντροφο, είπατε ότι θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Πιστεύω ότι πολλές από τις γυναίκες που μένουν μόνες τους, κυρίως τους ε, συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο παιδιά τους, στην επαγγελματική τους δραστηριότητα κρατάνε για αυτά την ενέργεια παρά να επενδύσουν στο να βρουν ένα νέο σύντροφο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ματήρα και κατόπιν ε, η κυρία Μασέλα Κόρση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις, ε, τις προσκεκλημένες εμπειρογνώμονες για όλα αυτά τα στοιχεία προσκέψη που μας δώσανε σε θέματα που καθημερινά συζητάμε στην Επιτροπή μας για τις ίσες ευκαιρίες αλλά και άλλα στοιχεία που ό,τι βλέπω είναι νέα επιπλέον και θα μας βοηθήσουν να μελετήσουμε και άλλα θέματα στο μέλλον. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Ευχαριστώ την καθηγήτρια Σάντα Μολίν και για τη μεγάλη εμπειρία της και από την Ιταλία και από την Ευρώπη σε θέματα ίσων ευκαιριών και πολιτικές συμφιλίωσης μεταξύ οικογένειας και επαγγελματικής ζωής. Την ερωτώ ποια στρατηγική, ποια μέθοδο έρευνας μας συνιστά για το μέλλον, για το μέλλον. Και προς την καθηγήτρια ερωτώ ποια είναι η γνώμη σας να έχουμε έναν χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της γυναίκας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο χρόνος αγορεύσης είναι ένα λεπτό μόνο για να προλάβουμε να ακούσουμε τους πάντες. Και κάντε ερωτήσεις παρακαλώ, όχι δηλώσεις. Η καθηγήτρια μας έλαγκώσει τώρα. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ανάλυσης των θεμάτων των φύλων σε σχέση με την πολλοπηγή άνηση μεταχείριση. Αυτό είναι σημαντικό. Ταυτόχρονα όμω, θα πρέπει να μετρήσουμε το τι έχει γίνει ήδη. Και όσον αφορά δείκτες ad hoc που είναι σημαντικοί Βέβαια, μια ομάδα η οποία έχει επιφορτιστεί με το θέμα αυτό ακόμα δεν έχει φέρει σε πέρας το έργο της. Κυρίως όμως πρέπει να δούμε το ρόλο των γυναικών στην οικογένεια με δείκτες και με παραμέτρους, ενισχύοντας τις στατιστικές πηγές που έχουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο μία συγκεκριμένη database, δεν αρκεί όμως. Έπειτα οι common indicators που χρησιμοποιούνται από την κοινότητα δεν χρησιμοποιούνται 100% ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ διαφόρων οικογενειακών πυρήνων που όπως είδαμε από τις σημερινές παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της επίπτωσης της πολιτικής για τους άντρες και τις γυναίκες. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βίκη Κλίζα από το EPPF. Okay, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το IPPF έχει συμβάλει στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Και μετά όπως ακούστηκαν από τις ομιλητές, θα ήθελα να τονίσω και εγώ τρεις τομείς που δεν ε, εκπροσωπούνται πάρα πολύ ε, στην έκθεση και να θέσω ένα ερώτημα αν μπορούμε σε αυτούς τους τρεις τομείς να δράσουμε λίγο περισσότερο. Ένα είναι ο τομέας της υγείας, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία κυρίως, Ακούσαμε το πόσο σημαντικό είναι ο τομέας αυτό στη ζωή και το μέλλον μιας γυναίκας. Ο άλλος τομέας που θα ήθελα να θίξω είναι η βία εναντί των γυναικών. Ίσως θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό στα πλαίσια και των μελλοντικών στρατηγικών. Εκεί θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική εκπαίδευση, την κατάρτιση ε, κοριτσιών και αγοριών στο σεβασμό του ενός προς τον άλλον, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και τέλος, ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι θα λύσουμε τα πάντα, αλλά είναι ένα σημείο κλειδί. Και οι γυναίκε πρέπει να, να κάνουν δύο φορέ και τρει φορέ την ίδια προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τέτοιε καταστάσει και νομίζω ότι θα πρέπει να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Η Λουίσα Αντολίν. Δίκτυο Βίντεν, παρακαλώ. Καλημέρα. θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση κυρίως για την ε, νέα στρατηγική ως προς εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κατάλαβα καλά, η καθηγήτρια Walby είπε ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία και μετά άκουσα την παρέμβαση της κυρίας Πάικ και μου έδωσε εντύπωση ότι δεν μας μίλησε για νέα στοιχεία, ήταν λίγο ασαφής ε, στην παρουσίασή της. Ε, μας, μίλησε για, μας μίλησαν ε, διάφορες ομιλήτρες για ανακολουθίες ανάμεσα σε τμέρες πολιτικές της Ένωσης. Πάντως ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της ισότητας των δύο φύλων και όχι μόνο στο εσωτερικό της αλλά και στις σχέσεις της ε, με τρίτες ε, χώρες. Γιατί ξέρετε έχουμε και υπηκούς τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει απομόνωση, υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μεν και στις δε. Αλλά ε, πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε τα του οίκου μας. Αυτό το νέο σχέδιο δράσης ε, νομίζω θα πρέπει να έχει ισχυρή εξωτερική διάσταση. Από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Γυναικών, η κυρία Γκονζάλης τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την ε, δόκτωρα Τζοβάνα Νταμολίν το εξής. Θεωρείτε ότι αρμόζει να προσθέσετε κάποια στοιχεία, παραδείγματο χάρη, ε, πώ να μεταχειριζόμαστε τι ηλικιωμένε γυναίκε που δεν μπορούν να πάνε σε οίκο ευγυρία, ε, δεν τους το επιτρέπουν τα οικονομικά τους δηλαδή. Ποια στήριξη μπορούμε να ε, προσφέρουμε σε αυτές τις γυναίκες ε, για να ε, παραμείνουν στο σπίτι τους έχοντας κάποια φροντίδα. Δεύτερον, πώς πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες που περιθάλπουν τους ηλικιωμένους. Δηλαδή πώς να αναγνωριστούν οι περίοδοι, ο χρόνος ε, που ε, δαπανούν για αυτή την φροντίδα με φορολογικά κίνητρα. Τρίτον, ε, υπάρχουν γυναίκες που ε, επειδή πρέπει να περιθάλψουν οι ηλικιωμένους ε, με ηλικογενεία, σε ανάπηρα παιδιά πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους. Ε, ποια βοήθεια μπορούμε να τους δώσουμε και τέλος η συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής κρίνεται. Ότι θα πρέπει να προβλέπετε για προσωπικούς λόγους η δυνατότητα σας και στις γυναίκες να παραμένουν μεγαλύτερο χρόνο στο σπίτι τους. Σας ευχαριστούμε όλους για τις ερωτήσεις σας. Θα έχετε και πάλι τη δυνατότητα να ε, υποβάλλετε ερωτήσεις μετά το επόμενο πάνελ, την επόμενη ομάδα συζητήσεων. Τώρα θα ήθελα να μας ε, απαντήσουν ε, οι προσκεκλημένες μας σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άπειρο χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, θα ορίσω το χρόνο των απαντήσεων στα τρία λεπτά λοιπόν. Α, και η κυρία Πάικ πρέπει να απαντήσει στη συνέχεια. Η κυρία Βάλμπη θα πάρει πρώτη το λόγο. Μάλιστα. Ε, με ρώτησαν ε, ε, πολύ για τα ανθρωπίνα δικαιώματα, για αυτό το χάρτη που προτείνει ο πρόεδρος Μπαρόσο. Το θέμα των δικαιωμάτων, τα θέματα δικαιώματων αναπαραγωγής, διάφορες ερωτήσεις. Λοιπόν, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει ισχυρή τάση αλλά δεν έχει θεσμοποιηθεί το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης επαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, έχει πλεονεκτήματα, έχει και ατέλειες. Αναγνωρίζεται η βία ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ και το ίδιο ισχύει και για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Σε διεθνές επίπεδο ήρθε η ώρα να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση των ΟΗΕ κατά ε, τον ΙΠΑ για τα θέματα αναπαραγωγικών δικαιωμάτων ε, με τη νέα κυβέρνηση στη ΣΥΠΑ πρέπει να έχουν επιλογή οι γυναίκες για την άμβλωση. Πρέπει να εγγραφεί στην, μερίσια, διεθνή, διάτα, στην Διεθνή Μερίσια Διάταξη και πάλι το ζήτημα. Έχουν πει οι ότι σκοπεύουν να αλλάξουν τη θέση τους, λοιπόν να πιέσει η Ένωση για το θέμα των δικαιωμάτων ε, σεξουαλικής ε, ζωής και αναπαραγωγής. μπορούμε να έχουμε νέες ε, παρεμβάσεις ε, και το θέμα τώρα της διατομιακής συνεργασίας ανάμεσα στα ιδρύματα, ναι, έχετε δίκιο. Ε, βλέπουμε συγχώνευση ε, των εθνικών Ινστιτούτων και σε όλα αυτά τα σημεία που έγινε συγχώνευση αποδυναμώνεται αυτή η συνιστόσα της προστασίας των, ε, της ισότητας των δύο φύλων. Δεν φταίει η ίδια η συγχώνευση. Είναι που δεν αναδεικνύεται σε βασική πολιτική το θέμα της προστασίας. Μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα να αναλύσουμε την κατάσταση για να δούμε τι χάθηκε, τι έγινε. Πριν τη συγχώνευση των Ινστιτούτων, τα Παλιά οι ε, ε, ε, Ινστιτούτα είχαν ασχοληθεί με διάφορα ζητήματα, φιλετικά και άλλα. Δεν νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε. Τώρα με το νέο μηχανισμό που έχουμε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ισχυρές παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε η κυρία Νταμολίν. Grazie per questi interventi che richiamano l'attenzione sulle questioni demografiche soprattutto. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ότι αναφέρατε τα δημογραφικά προβλήματα. Αρκετοί από εσά αναφέρθηκαν στα δημογραφικά προβλήματα και στις ηλικιωμένε γυναίκες. Αυτό όντω είναι κάτι που μετατρέπεται σε απειλή για το μέλλον και χρειάζεται την προσοχή μας stiamo lavorando anche come demografe. Eh, Μιλώ για, στην έκθεσή μου για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες αυτές για υποκατάστατα περίθαλψης, καθώς επίσης για οικιακή βοήθεια, βοήθεια στο σπίτι. Νομίζω ότι επ' θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα χρόνια που έρχονται. Ένα άλλο που ήθελα να θίξω ήταν ε, οι χωρισμένες γυναίκες και οι εργένισες. Δεν ε, ήθελα να πω ότι όλες θα πρέπει να βγουν και να αρχίσουν να ψάχνουν για σύντροφο, αλλά ε, ίσως να υπάρξει μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα παραμείνουν μόνες τους και μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν ε, και τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να είναι και μεταβατικό στάδιο στη ζωή τους, αλλά είναι αρκετά επικίνδυνο. Γιατί αυτές οι γυναίκες είναι μόνες τους, δεν έχουν ε, σύζυγο ή σύντροφο, οπότε ίσως όντως να είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια βοήθεια. ίσως να υπάρξει κάποια οικονομική ενίσχυση μέχρι να ξαναγίνουν μια φυσιολογική οικογένεια. Αυτό εννοούσα, ότι θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια για τις γυναίκες αυτές κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που είναι μόνες τους. Ε, Μόλις γυναίκες βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να τους, υπο... να τους δίδεται και βοήθεια. Και τέλος, το πρόβλημα που ανέφερε η καθηγήτρια Ματέρα. Νέα μεθοδολογία για την έρευνα. Ακούσαμε ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία κατά φύλλο, άρα χρειάζονται τράπεζες δεδομένων επίσημες να υπάρξουν δείκτες και παράμετροι ομοιογενείς δείκτες ελέγξιμοι που να ισχύουν για όλη την Ένωση ομοιόμορφα και προσθέτω νέες έρευνες επιτόπια να ακούσουμε τις γυναίκες η πολιτική να μην είναι μια υπερδομή οι επιλογές να γίνονται από τις γυναίκες οι έρευνες, κοινωνικές έρευνες να γίνονται επιτόπου με focus groups και λοιπά, να ακούσουμε τις γυναίκες τι έχουν να πούνε για τη ζωή τους. Και από εκεί να απορρέει η πολιτική, μετά από τις γυναίκες. Ένα είδος διαβούλευση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρίσα Σολέτο. Σε πέντε και τρία λεπτά τώρα να απαντήσω και μεγάλη ευχαρίστηση όλα όσα υπόθηκαν. Θα αναφερθώ σε τρία θεμελιώδη σημεία. Διεθνείς σχέσεις. Επίγει τα όργανα και οι γυναίκες στις αναπτυγμένες χώρες να ξέρουμε να έχουμε επίγνωση της ευθύνη μας και να απαιτήσουμε από τις χώρες μας να ενσωματωθούν οι προτεραιότητες για τα δικαιώματα των γυναικών σε θέματα διεθνών σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας η Ένωση θα πρέπει να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του, της απόφασης 1325 του Συμβουλίου γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη μηχανισμούς σχετικούς μιλάμε για πράξεις, πολλές, δράσεις συγγνώμη, πολλές φορές κοινέ. συλλογική δράση το, διότι απαιτούνται οργανισμοί σε πολλά επίπεδα που να δουλεύουν συντονισμένα με συγκεκριμένα κονδύλια και προπολογισμό και για κάθε δράση να υπάρχουν άτομα υπεύθυνα για την ισότητα και να υπάρχουν και άτομα για τον συντονισμό. Αν αυτά τα δύο επίπεδα θεσμικής δράσης δεν τα έχουμε, τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Το ξέρουμε αυτό. Οι επιπτώσεις, οι θετικές επιπτώσεις στην πολιτική θα χαθούν. Όποια ανάγκη λοιπόν και να γίνει αυτά τα δύο επίπεδα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς κατά νου. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στη διαφορά από την θέση που έχω επειδή έχω συνεργαστεί με άτομα που δουλεύουν για την, κατά της άγγισης μεταχείρισης το θέμα των φύλων στη διάκριση είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και χρειάζεται πολλή δουλειά για να εντοπιστεί ότι το φύλλο είναι πολύ σημαντικό το θέμα του φίλου και δημιουργεί νέες καταστάσεις όταν συνεργαζόμαστε με άλλους που ασχολούνται με το θέμα της διαφοράς ή των διαφορών. Το θέμα του φύλου, δηλαδή οι γυναίκες υπήρχε η των διαφορων το θεμα του φιλου δηλαδη κατά της ανήσης μεταχείρισης με βάση την ε, εθνοτική προέλευση κλπ. κλπ. Τώρα, αν δούμε τα θέματα ισότητα για όλους, το δικαίωμα στη διαφορά, πρέπει να το δούμε διαφορετικά και με πολύ πιο σοβαρό τρόπο. Και τέλος, η συμμετοχή των ανδρών είναι να μοιράζεται η δουλειά. Να μοιράζεται η δουλειά μεταξύ ανδρών και γυναικών και στο σπίτι. Μπορεί να υπάρξουν νομοθεσία που να ε, ε, δίνουν κίνητρα στον άντρα να λάβει και αυτό το έργο μέσα στην οικογένεια. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πάικ γιατί σας ρώτησαν κάτι για, τη δημογραφική, για τις δημογραφικές εξελίξεις και την πληθυσμιακή γύρανση. Ναι, ούτως ή άλλως θα μιλήσω και αργότερα. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις θα κάνω. Βέβαια, το δημογραφικό πλαίσιο ορίζει οτιδήποτε αποφασίσουμε στα πλαίσια της στρατηγικής και αυτό πρέπει να είναι σαφές ε, στα πλαίσια της νέας στρατηγικής, αλλά η οτιδήποτε κάνουμε επίση για τι ε, συντάξεις ή οποιαδήποτε απάντηση δίνουμε στι δημογραφικέ τάσει, ε, πρέπει να ε, βασίζεται στην κατανόηση των διαφορών που υπάρχουν και των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλλα. Επίσης είπαμε πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα σε διάφορου τομεί, αλλά μην υποτιμάτε αυτά που ήδη υπάρχουν γιατί δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε ικανοποιητικά ακόμη και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες μπορούν να κινηθούν ούτως ώστε να έχουμε δεδομένα σε διάφορους τομείς και τα χρησιμοποιήσαμε για τις εκθέσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πριν από τα Χριστούγεννα που σας ε, μοιράσαμε. Είναι στο παράρτημα της έκθεσης και τα δεδομένα δείχνουν ότι συμβαίνει στα κράτη-μέλη σε διάφορους τομείς. Ο κίνδυνος για τη φτώχεια, παραδείγματος χάρη. Βλέπετε σε διάφορες χώρες, στη Σλοβενία, στη Βουλγαρία, αλλά και σε άλλες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία και Ρουμανία, οι γυναίκες άνω των 65 έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας σε σχέση με τους άντρες. Χρειαζόμαστε δεδομένα για να στηρίξουμε τη δουλειά μας. Για το ρόλο των αντρών τώρα κάναμε με το Αυροβαρόμετρο μία δημοσκόπηση. Θα δημοσιευθούν σύντομα τα αποτελέσματα και το ενδιαφέρον ήταν ότι Κάναμε διάφορε διαπιστώσει. Ο, αν έχει υψηλότερο εισόδημα η γυναίκα, πρέπει να μείνει ο άντρα στο σπίτι και να φροντίζει τα παιδιά. Η το ποσοστό γυναικών πιστεύουν πως όχι παραδόξως. Ε, πρέπει να πηγαίνει ο άντρας να δουλεύει. Ε, άρα ε, επίσης για την ανατροφή των παιδιών, ναι. Ένα, μας ξαφνιάζει πόσο υψηλό είναι το ποσοστό των γυναικών που πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να μένουν στο σπίτι να φροντίζουν τα παιδιά. Είναι περίπλοκη, περίπλοκο το φαινόμενο παρότι έτσι ε, ε, σας μιλάω για περιπτώσεις όπου είναι υψηλότερο το εισόδημα της γυναίκας η γυναίκα και ο άντρας πρέπει να είναι σύμμαχοι ε, γιατί τα ίδια στερεότυπα που παγιδεύουν τις γυναίκες παγιδεύουν και τους άντρες για την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας. Φυσικά ασκούμε τις εξουσίες που έχουμε τόσο ώστε να μεταφέρονται σωστά ε, τα νομοθετήματα στην εθνική νομοθεσία αλλά το άλλο θέμα είναι πώς ακριβώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται μέσα στην νομοθεσία και έχουμε και εδώ το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ενημερώνουν του πολίτες πολίτε, ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώ να τα εφαρμόσουν. Και αυτό θα μας απασχολήσει, ούτως ώστε ένα υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού να γνωρίζει τα δικαιώματά του. Επίσης για τα δικαιώματα μην ξεχνάτε ότι έχουμε σημαντικό όγκο ε, κοινοτικών νομοθετημάτων για τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Ε, έχουμε και τις διεθνεί συμβάσει, τη Διεθνή Σύμβαση ΙΝΤΟ και ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα βελτιώθηκε η κατάσταση με τη νέα συνθήκη. Οπότε το θέμα είναι πώς να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία. Αν χρειάζεται κάπου νέα νομοθεσία, εντάξει, ας το εξετάσουμε, αλλά Α ε, τονιστεί η σημασία της εφαρμογή της ήδη υφιστάμενης νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Πάικ. Ευχαριστούμε τις ομιλήτριες της πρώτης ομάδας. Συνέβαλαν ουσιαστικά αυξάνοντας τις γνώσεις μας για το θέμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ένα θερμό ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ακρόασή μας και πριν καλωσορίζω τα μέλη της δεύτερης ομάδας ε, θα ήθελα να σας πω και κάποια πράγματα. Ε, διάφορες ομιλήτρες ε, ήταν ταχύτατες και δυσκολεύονται οι να παρακολουθήσουν. Οπότε ήθελα να το έχετε κατά νου. Σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά. Δεύτερον, ε, μου είπε κάποιος ότι σε διάφορες ε, γλώσσες δεν μεταφράζεται η λέξη πρόεδρος στο θηλυκό του. Ο ή πρόεδρος στα ελληνικά δεν τίθεται το ζήτημα. Θα συζητήσουμε τώρα για τα μέσα και για τα εργαλεία για μια αποτελεσματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη από όλους θα μιλήσει η κυρία Μύρια Βασιλιάδου που είναι Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών. Καλώς ορίσατε. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Γυναικών που προσκάλεσε το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών. Έχουμε ακρά αγώνιμη συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρόεδρο που μας προσκάλεσε. Και έχουμε συνεργαστεί με πολλούς ε, επιμέρους ευρωβουλευτές, άνδρες και γυναίκες από όλα τα πολιτικά κόμματα που μας βοήθησαν ιδιαίτερα στην τελευταία καμπάνια, οι γυναίκες και οι αποφάσεις. Ήδη αναφέρθηκε ότι μπροστά μας έχουμε προκλήσεις. Financial and Έχουμε την, κράση, την κρίση, την οικονομική κρίση, Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας που άρχισε να ισχύει. Έχουμε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπό τον νέο επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά στη δουλειά μου. I will just say a slide of who we are to remind those of you who might not uh, remember or are not familiar. Καταρχήν σας θυμίσω ποιοι είμαστε και θα σας μιλήσω για τον οδικό χάρτη, για τις προκλήσεις και κυρίως συστάσεις για το μέλλον. Πρώτον, είμαστε πιο μεγάλη οργάνωση ομπρέλα για την Ένωση των Γυναικών στην Ένωση. Έχουμε εθνικούς συντονιστές σε όλα τα κράτη-μέλη και ασχολούμαστε με την πολιτική δουλειά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το ερώτημα από τον ειδικό χάρτη, θα αναβερθώ κυρίως στην διαβούλευση που υποβάλαμε στην Κομισιόν, στην Επιτροπή για τον μελλοντικό οδικό χάρτη στην είσοδο της έδωσας υπάρχουν φάκελοι σχετικά με το θέμα αυτό. Τι ζητήσαμε από την Επιτροπή. Επίσης, ασχολούμαστε με τη γνωμοδότηση που βγήκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν για τις ίσες ευκαιρίες ανδρών γυναικών εκεί το λέγειν το έχουν οι χώρες μέλη. Για τον οδικό χάρτη επανέρχομαι. Υπόθηκαν ήδη αρκετά. Να σας αναφέρω κατά λέξη τι υποβάλαμε στην Κομισιόν. Ο οδικός χάρτης ήταν περισσότερο ένας εσωτερικός συντονιστικός μηχανισμός για την Επιτροπή παρά ένα δεσμευτικό έγγραφο πολιτικής και στηρίζεται κυρίως σε προαιρετικό input εκ μέρους των υπηρεσιών της Κομισιόν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς λέμε, χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό πρόγραμμα δράσης για πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών με συγκεκριμένα μέτρα και μηχανισμούς απόδοσης ευθύνης. Και ευχαριστούμε την κυρία Πάικ που έκανε ένα θετικό επινιγμό στο θέμα αυτό. Τα θετικά στοιχεία του οδικού χάρτη αναφέρονται και στις συγκεκριμένες δράσεις και στο γενικότερο mainstreaming. Αφορά την ισότητα σε, όλες, σε όλα τα επίπεδα ζωής και έχει προτεραιότητες πέραν πέραν των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικές όπως η βία κατά των γυναικών, οι γυναίκες και οι αποφάσεις, εκπαίδευση, ανάπτυξη, συνεργασία κλπ. Θα επανέλθω σε αυτό. Η πρώτη πρόκληση που ήδη αναφέρθηκε αναφέρεται στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Έχουμε ένα σύστημα που σε μεγάλο βαθμό απέδειξε ότι απέτυχε. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία της κρίσης να κάνουμε κάτι άλλο, ένα διαφορετικό μοντέλο προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε προγράμματα ανάκαμψης με αξιολόγηση των επιπτώσεων μικρών γυναικών. Το σχέδιο της Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν το εμπεριέχει αυτό. Πρέπει να δούμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η δημόσια δαπάνη για τις γυναίκες. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περίθαλψη. Περίθαλψη για τα παιδιά, αλλά η περίθαλψη ευρύτερα. Για τους ηλικιωμένους και βαθιά επανέλθει και σε αυτό. Ήδη κάναμε μια δήλωση και συστάσεις οι γυναίκες και η κρίση και κάνουμε έρευνα με την Oxfam για τις επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες. Μιλάμε, αλλά συγκεκριμένα αποτελέσματα ακόμα δεν έχουμε. Τη λέμε η άδειλη κρίση, μη εμφανής κρίση. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε η καθηγήτρια Γόλμπη η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένας στόχος. Τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον ακούμε ότι χρειαζόμαστε ισότητα γιατί χρειαζόμαστε απασχόληση, οικονομική ανάπτυξη κλπ. Χρειαζόμαστε ισότητα για την ισότητα. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό όταν μιλάμε για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και για το στρατηγικό σχέδιο. Δεν είναι απλώς επαγγέλματα, απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε επίση συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου. Κάτι άλλο που χαίρομαι που το ανάφεραν οι ευρωβουλευτέ, είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν πρέπει να χάνεται με τη συζήτηση ισότητα για όλου. Σαν είναι δευτερεύον το θέμα δηλαδή της ισότητας των φίλων και έχουμε και τις προτάσεις της Κομισιόν για την κατά της άγγισης μεταχείρισης που την υποστηρίζουμε αλλά ταυτόχρονα κρούμε τον κόδωνο του κινδύνου και για τους ευρωβουλευτές για το ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην ομοθεσία σχετικά με τα φύλλα και αν αυτή η πρόταση κατά της άγγισης μεταχείρισης δεν έχει μέσα μια ισχυρή συνιστόσα mainstreaming θα έχει αποτύχει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι θετικό το ότι η Ισπανική Προεδρία το φέρει πάνω στο κέντρο η βία κατά των γυναικών και υπάρχει ανάγκη για νομική βάση γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι και επαρκής προστασία της ε, αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών και τι γίνεται στα Ηνωμένα Έθνη και να δούμε στην εξωτερική μας πολιτική και την ιστορική πολιτική μήπως υπάρχουν αντιφάσεις για τα δικαιώματα αυτά και να φέρουμε υποχρεωτική στήρωση, πρόσβαση στη μητρική φροντίδα, σε φροντίδα για τις έγκυες οι νόμιμες ε, εκτρώσεις όπου αυτό ε, επιβάλλεται κλπ. Στρατηγικό πρόγραμμα δράσης. Εδώ το πιο σημαντικό είναι η ανάγκη να είμαστε προδραστικοί. Γιατί η ισότητα των φίλων δεν είναι απλώς δράση κατά της άγγισης μεταχείρισης. Μπορεί να έχετε ό,τι θέλετε κατά της άγγισης μεταχείρισης χωρίς να έχετε ισότητα. Και η βία που στηρίζεται στα φύλλα το βλέπουμε, είναι το καυτό σημείο. όσον αφορά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους πολλά υπόθηκαν να χρειαζόμαστε δομές προκειμένου να πετύχουμε την ισότητα των φύλων μέσα στα πλαίσια περικοπών που ζούμε και χρειάζεται και ένα συντονιστικό φορέα που σημαίνει το προσωπικό που δουλεύει για το mainstreaming πρέπει να είναι εμπειρογνώμονε, να έχουν πόρου για κονδύλια, να είναι εμφανεί να μην άτομα που έρχονται και παρέρχονται, όπως συνήθως συμβαίνει, συνήθως σε επίπεδα κρατών μελών ή και σε ευρωπαϊκό, κάνουμε και λίγο mainstreaming ή ελάτε στην Επιτροπή για λίγο χρονικό διάστημα και φύγετε. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Σε σχέση με το στρατηγικό σχεδιασμό, χρειαζόμαστε συγκεκριμένη δράση, χρειαζόμαστε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, και πρέπει να δούμε τους έξι τομείς του οδικού χάρτη και έχουμε συγκεκριμένες συστάσεις από αυτού Επιπλέον όμως πρέπει να εστιαστούμε στη βία κατά των γυναικών δεσμευτικά μέτρα αυτό να δούμε τη νομική βάση πριν να πούμε κάτι για τη μετανάστευση, την ασωμάτωση και το άσυλο, που γίνεται όλο και πιο επίκαιρο θέμα, όπως επίσης αυτό που ήδη συζήτησαν οι βουλευτές σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και το θέμα της υγείας. Θα προσπαθήσω να τελειώσω σε ένα λεπτό. Το θέμα αυτό της διτής προσέγγισης, στην οποία αναφέρεται η Μπελίντα Πάικ, πρέπει να συνεχιστεί και οι ειδικέ δράσεις οπωσδήποτε δεν πρέπει να πάψουν να εφαρμόζονται. αυτό είναι μια τάση ε, την οποία πρέπει να καταπολεμηθεί, πρέπει να σταματήσει. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο έγγραφό μας σχετικά με τους στόχους και τους δείκτες. Θέλουμε να τονιστεί το θέμα της περίθαλψης για τους εξα... εξατόμενα άτομα όλων των ηλικιών και όλων των ομάδων, γιατί υπάρχουν τεράστια κενά σε αυτό και τελειώνω και λυπάμαι που ήμουν υποχρεωμένη να είμαι αρκετά συνοπτική επειδή δεν έχω χρόνο θέλουμε την πλήρη εφαρμογή του, των πλαισίων για την ισότητα των φύλων. Δεν το έχουμε. Έχουμε το ΣΥΝΤΑΛ, το Πεκίνο και τα κράτη-μέλη τα έχουν υπογράψει όλα αυτά. Αυτό που θέλουμε είναι επιπλέον μέτρα και τρόποι για να εφαρμοστούν αυτά. Έχουμε το ΣΥΝΤΟ. Καλό είναι το ΣΥΝΤΟ, αλλά δεν εφαρμόζεται από τις περισσότερες χώρες μέλη. Καλούμε τις κυβερνήσει να φροντίσουμε κάτι να γίνει και γι' αυτό. Και μια διάσταση για το φύλλο να μπει στη στρατηγική του 2020 έχουμε την ετήσια έκθεση της Κομισιόν ψηφωνούμε κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό δεν τα είπα όλα όσα ήθελα να πω ευχαριστώ που με ακούσατε Ευχαριστώ. Λυπάμαι πραγματικά που δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα που μας απασχολούν. Πάντως σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα περάσουμε στην κυρία Οντέτ Φιλίπε, που είναι συντονιστρία στην Επιτροπή ε, Ισότητας της Γενικής Συνομοσπονδίας Πορτογάλων Εργαζομένων. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή σας. Μπορώ να έχω τη δυνατότητα να έρθω να σας παρουσιάσω όχι μόνο την κατάσταση στην Πορτογαλία, να κάνω και κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της κοινωτική πολιτικής και να μάθω πράγματα από εσά βέβαια. Θα ήθελα να περιγράψω σύντομα την κατάσταση στην Πορτογαλία. Λοιπόν, οι εργαζόμενες μετά από την επανάσταση 25 Απριλίου του 1974 κατοχύρωσαν τα δικαιώματά τους στο Σύνταγμα και στην Εθνική Νομοθεσία. Ισότητα λοιπόν στη μεταχείριση, ισότητα στα δικαιώματα και ισότητα στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια, όμως σημειώθηκε μεγάλη οπισθοδρόμηση γιατί δεν, δεν εφαρμόζεται ούτε η εθνική ούτε η διεθνή ομοθεσία σωστά και υπάρχει σοβαρή οικονομική κρίση που πλήγει τις πλέον ευαίσθητες, ας το πούμε έτσι, πληθυσμιακές ομάδες. Οπότε ε, η ανεργία είναι υψηλότερη στις γυναίκες, επισφαλείς θέσεις εργασίας, χαμηλή μισθή, χαμηλές συντάξεις, ανισότητες, ε, διακρίσεις, ε, φτώχεια, χαμηλή πρόσβαση στι κοινωνικές υπηρεσίες υπηρεσίες πρόνοιας. Η μητρότητα παρά την νομοθεσία που τους προστατεύει δεν προστατεύεται επαρκώς ούτε στο χώρο εργασίας ούτε ως προς την προστασία της οικογενειακής ζωής και άρα η συμφιλίωση της οικογενειακής επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής δεν είναι ικανοποιητική. Δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες ε, ε, διαβίωσης. Ε, το 47% του δυναμικού είναι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Έχουν υψηλότερη μόρφωση συνήθως από τους άντρες. Παρόλα αυτά στο τρίτο τετράμινο το 2006 ήταν 10,6% το ποσοστό της ανεργίας, ενώ για τους άντρες ήταν 9,1%. 58,3% των εργαζομένων ε, μέχρι ανάμεσα ε, στα 25 ε, και από 25 μέχρι 33 ετών δεν έχουν μόνιμη σύμβαση εργασίας. Ο μέσος μισθός είναι χαμηλότερος σε σχέση με των γυναικών κατά 6%. Η προσφορά ε, θέσεων στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένες ε, θέσεις ε, δεν παρουσιάζει μία διαφορά 30% ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες και ο κατώτερος ο μισθός στην Πορτογαλία προς το παρόν είναι 450 ευρώ και υπάρχουν 20% των γυναικών που παίρνουν αυτό το κατώτερο μισθό ενώ για τους άντρες το ποσοστό είναι 5%. Επίσης, ε, στις παροχές για τη μητρότητα και για την πατρότητα, για, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες. Το 2009 η σύνταξη των γυναικών σε μέσο όρο αντιστοιχούσε στο 60% της αντίστοιχης σύνταξης για τους ε, άντρες. Αλλά ε, σε σχέση με την απασχόληση και με τους μισθούς πλήγονται ιδιαίτερα οι γυναίκες λόγω των ε, αρνητικών εξελίξεων στις επιχειρήσεις επειδή δεν ισχύουν πλέον συλλογικές συμβάσεις, οργανώνουν τη εργασία με νέους, με τρόπους παρατείνονται τα ωράρια εργασίας ε, και αυτό συνεπάγεται νέα προβλήματα για την υγεία και αναταράσσουν την οικογενειακή και προσωπική ζωή. Κάθε φο... Ε, ολένα και περισσότερο λόγω του εντατικού ρυθμού εργασίας υπάρχουν σοβαρές επαγγελματικές ασθένειες στις γυναίκες ε, και όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις, όταν υπάρχουν μαζικές απολύσεις, τελικά οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να βρουν νέα θέση εργασίας. Ε, τώρα, 12 ε, ώρες ε, την ημέρα δουλεύουν οι γυναίκες για να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ούτε αύξηση του μισθού, ούτε υπερορίες αναγνωρίζονται και αυτό αποτελεί παραβία των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών και θα ήθελα να τονίσω ότι οι δομές υποστήριξης ε, της οικογενειακής ε, ζωής ε, είναι ανεπαρκής γιατί πέρα από την κανονική δουλειά τους οι γυναίκες πρέπει να περνάνε ατελείωτες ώρες στο σπίτι για την προστασία των, συγγνώμη, για την φροντίδα των παιδιών και την περίθαλψη των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια. Οπότε πώς μπορεί να επλακεί όλη η κοινωνία, όλοι οι εργαζόμενοι, όλες οι εργαζόμενες στον αγώνα για την ισότητα ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη, καλύτερη συμπερίληψη όλων στην κοινωνία και να είναι πιο δημοκρατική η κοινωνία μα. μας. Ε, οι εργοδότε θα αναγνωρίζουν την κοινωνική αξία και τη μητρότητα και τη πατρότητα και να σεβαστούν τα δικαιώματα όλων. Τι να κάνουμε, ούτω ώστε η εργασία των γυναικών να αναγνωριστεί και να αμείβεται δίκαια και να ε, πλαισιώνεται σωστά μέσα από τι συλλογικέ συμβάσει, ε, Από τη δική μου εμπειρία, γιατί είμαι και συνδικαλίστρια και συντονίστρια τη Επιτροπή για την Ισότητα στην Πορτογαλική Συνομοσπονδία, θα ήθελα να προτείνω τα αποτελέσματα των εργασιών μα. Παρεμβαίνουμε στου χώρου εργασίας για την καταπολέμηση των διακριτικών ε, μεταχειρήσεων. Επεμβαίνουμε σε συγκεκριμένε καταστάσει, κάνουμε ενημερωτικέ εκστρατείε, ευαισθητοποιούμε ε, το κοινό ω προ τα δικαιώματα των γυναικών και προωθούμε την αξία των συλλογικών συμβάσεων. Ενισχύουμε τις ε, τοπικέ δράσει που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και προσπαθούμε να αναπτύξουμε μία αναλυτική μεθοδολογία για να προάγουμε την αξία της εργασίας ε, χωρίς διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα, ε, ε, απηχώντας έτσι την σχετική σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σχετικά με την ισότητα στον χώρο εργασίας και την, τις ίσες αμοιβές θα ήθελα να τονίσω ότι χάρη στις εργασίες μας από τον Ιανουάριο υπάρχει και μια σχετική κατάρτιση που προσφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας για τα ζητήματα που μας απασχολούν. Υπάρχουν δυνατότητες παρά τις δυσκολίες που σημειώνονται και θέλω να τονίσω εδώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προσδιοριστούν οι πολιτικές και να κινητοποιηθούν τα μέσα ούτω ώστε να ε, ε, ε, υλοποιηθεί η ισότητα ω προ τα δικαιώματα και να εναρμονιστούν οι διατάξει για να μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα προγράμματα στον τομέα τη ισότητας των δύο φύλων θα πρέπει να αποσκοπούν στην ανάληψη νέων δραστηριοτήτων για την προστασία των γυναικών στον χώρο εργασίας και επίσης στον τομέα των κρατικών υπηρεσιών αλλά και στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να καταργηθούν όλες οι μορφές διακριτικής μεταχείριση άμεση και επίση, επίσης. Σεβασμός της αρχής της συμφιλίωση τη οικογένειακή και τη επαγγελματική ζωή, προσδιορίζονται σωστά τα ωράρια εργασίας και ορισμός ανώτατων ορίων διάρκειας που να μην επιφέρουν προβλήματα υγείας στους εργαζομένους επίσης. Ε, Εκστρατείε ενημερωτικέ ε, και διάδοση ε, πληροφοριών για τα δικαιώματα, κυρίω ω προς τη μητρότητα και στην πατρότητα, για να αλλάξουν οι νοοτροπίε και για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανισοτήτων ανάμεσα στου άντρε και στι γυναίκε. Μα ο κόσμος συναποτελείται από άντρε και γυναίκε. και άρα πρέπει να ισχύει η δικαιοσύνη και η ισότητα και για του δύο. Αν θέλουμε να μιλάμε για την ωραία Ευρώπη της ισότητας, ε, λοιπόν στην καθημερινή ζωή θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Och ehm, eh, ευχαριστούμε. Η κυρία Βεσέλα Καρα... Καραϊβάνοβα τώρα, α, αναπληρώτρια διοικητής του NSSI, Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης Βουλγαρία. Σας παρακαλούμε να μιλάτε αργά, λίγο πιο αργά. Δεν γίνεται οι δερμηνείς να σας μεταφράσουν σε αυτούς τους ρυθμούς. Радвам се и за мен е удоволствие и чест да имам възможността да изложа пред всички вас. Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα για να σας περιγράψω την κατάσταση στη δική μου χώρα στη φορά, την ε, ισότητα των δύο φύλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παρβάνοβα για την ε, πρόσκληση. Η Κομισιόν ε, έχει χαρακτηρίσει το έτος αυτό πολύ σημαντικό για την ε, ισότητα των δύο φύλων. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη και να σας δώσω έτσι κάποιες αδρές γραμμές της ε, Βουλγαρίας σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και τις στρατηγικές που ακολουθεί για τη βελτίωση της ισότητας των δύο φύλων. Και βεβαίως ό,τι θέλετε είμαι εδώ για να σας ε, απαντήσω. Πώς έχουν τα πράγματα. Βλέπετε εδώ στην οθόνη το νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς ε, δεσμεύσεις ε, τις οποίες ε, τηρεί η Βουλγαρία και επί τη βάση των οποίων έχει εκπονήσει την εθνική της στρατηγική. Το Σύνταγμα παραθέτει εδάφια με την με, την, με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των δύο φύλων, κοινωνική βοήθεια, κοινωνικό ε, κώδικα ασφάλεια, υπάρχει ο το εργασιακό, εργατικό δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο τη ε, απασχόληση, ε, κοινωνική βοήθεια, υπάρχει ο οικογενειακό κώδικα που παραθέτουν ε, αρκετά στοιχεία για την ισότητα των δύο φύλων. και υπάρχουν επίσης και περιορισμοί οι διεθνείς τώρα Υπάρχουν περιορισμοί για όλους αυτούς τους φορείς Υπάρχουν και οι διεθνεί μα δεσμεύσεις Μπορώ να σας αναφέρω την συνθήκη του Άμστερνταμ, της νίκιας, τον Ευρωπαϊκό Δικοχάρτη για την ισότητα των δύο φύλων του 2006 έως 2010 και την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης. Σημειώστε ότι ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για μας είναι το βασικό πλαίσιο με το οποίο η Βουλγαρία εκπώνησε τα εθνικά της προγράμματα για την ισότητα των δύο φύλων. Ο κοινωνικός κώδικας είναι ένα ειδικό κομμάτι νομοθεσίας το οποίο προβλέπει την ε, υποχρεωτική φύση για την ε, κοινωνική ε, ασφάλεια και επίσης την ισότητα των δύο φύλων. Παρά το ότι υπάρχει και ειδικό και γενικό ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχουν ακόμη κάποια τμήματα της νομοθεσίας τα οποία δεν εγγυώνται επαρκώς την ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους τομείς της ε, ζωής. Οπότε έπρεπε και εμείς να δημιουργήσουμε μια εθνική στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων. Οι βασικές της αρχές είναι οι συγκεκριμένε που βλέπετε στην οθόνη. Ανθρώπινα δικαιώματα, ίσα δικαιώματα, ίση συμμετοχή και ίση πρόσβαση σε πόρους για άντρες και γυναίκες, ισόρροπη εκπροσώπηση φίλων στην λήψη αποφάσεων, εταιρική σχέση, έλεγχος και εποπτεία. Ο έλεγχος και η εποπτεία στην Βουλγαρία εμπίπτουν στα πλαίσια της Επιτροπής για την Διακριτική Μεταχείριση, της οποίας ο πρόεδρος βρίσκεται εδώ, είναι ο κύριος Κεμάλα Γιούμπ και δείχνει ότι η χώρα μου Όντω με την πολιτική της στοχεύει στην αντιμετώπιση της διακριτική μεταχείρισης και στην προώθηση της δημόσιας συζήτηση, του δημόσιου διαλόγου για την ισότητα των δύο φύλων. Όντω πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά τη διακριτική μεταχείριση ε, ανάλογα με το φύλο, γιατί εκεί ακόμη υπάρχει αρκετό πεδίο δράσης. Στρατηγική στόχη και τομείς δράσης οικονομικό τομέα, Επίτευξη των ε, στόχων της Λισαβόνας στον ε, τομέα της απασχόλησης. Απάλληψη των ε, διαφορών των, του χάσματος του μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ισότητα στο, των δύο φύλων στην επιχειρηματικότητα και στη γεωργία. Ισότητα στην κοινωνική, στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στην αντιμετώπιση της ένδυας συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, εφαρμογή, αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών, στην απασχόληση, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κοινωνικές υπηρεσίες για, τους, για τα παιδιά και τους ενήλικες, προώθηση στην ισότητα των δύο φύλων στην εξουσία και στις, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, απάλληψη της βίας ε, ανάλογα με το φύλλο και, την, ε, και το εμπόριο ανθρώπων και επίσης ε, ισότητα των δύο φύλων στο σύστημα ασφάλειας. Οι πολιτικές αυτές θα αλλάξουν τα στερεότυπα και τις νοοτροπίες, ειδικά αυτά τα πεπαλαιωμένα στερεότυπα τα οποία οδήγησαν τελικά σε αυτή την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων και που προβάλλονται από τα ΜΜΕ. Ω κοινωνία των πολιτών θα έπρεπε να έχουμε μηδενική ανοχή εναντί σεξιστικών ε, διαφημίσεων και άλλου τέτοιου είδους ε, συμπεριφορά των ε, ΜΜΕ η οποία υποβιβάζει τι γυναίκε. Ο εκλογικό νόμο επίση θα πρέπει να αλλάξει για να εγγυάται ποσοστώσεις για την ε, ε, ένταξη και γυναικών στην ε, δημόσια ζωή. Στην διαφάνεια αυτή προσπάθησα να αναλύσω την αντιστοιχεία αντρών και γυναικών στις, στους λίστες για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2009. 33% για τις γυναίκες και 67% για τους άντρες. Αλλά στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Παρά λοιπόν την ανισότητα στα ψηφοδέλτια, υπάρχει μια σχετική ισότητα στα, α, στα αποτελέσματα των κομμάτων. Ας πούμε το γκέρπ, το κυβερνητικό κόμμα, η συντηρητική επίση, ε, η κίνηση για τα δικαιώματα και την ελευθερία. Κάποια από αυτά τα κόμματα έχουν ε, βάλει ε, στις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων τους τις γυναίκες. Και αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για το πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Γιατί οι εκλογές και το πώς εκτιλήσονται οι εκλογές καταδεικνύει περίπτρανα ποιες είναι οι αξίες ενός πολιτικού κόμματος. Οι γυναίκες στο κοινοβούλιο θα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμες ώστε να προχωρήσει, να προωθηθεί το θέμα της ισότητας των δύο φύλων μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα αναθεωρήσουμε τον, τη στρατηγική μας για την ισότητα των δύο φύλων Και θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και για τη δική μου χώρα, αλλά πιστεύω και για όλα τα κράτη-μέλη. Δημιουργούμε μια, ε, συνολική, ένα συνολικό εθνικό μηχανισμό για ίσες ευκαιρίες μεταξύ αντρών και γυναικών τα πλαίσια της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκε από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες στο Πεκίνο το 1995. Οικονομική επίσης ε, υποστήριξη, οικονομικές εγγυήσει, ε, γιατί είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου για την ε, Ισότητα. Είναι φορέας της κυβέρνησης αυτό στην Βουλγαρία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, ε, υπό, να υπόκεινται σε κυρώσεις αν δεν εφαρμόζουν σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εθνική, τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας θα πρέπει να εισαγάγουν σε όλη την Ευρώπη την ιδέα της ε, γονικής άδειας. Στη δική μου τη χώρα αυτό συμβαίνει. Και δυνάμει του βουλγαρικού δικαίου οι άντρε μπορούν να πάρουν γονική άδεια άδεια πατρότητας, αλλά υπάρχει η γνωστή παράδοση και το γνωστό στερεότυπο. Οι άντρες ακόμη και αν έχουν το δικαίωμα να πάρουν άδεια ε, γονική, δεν την παίρνουν τις περισσότερες φορές και είναι οι γυναίκες αυτές που μένουν σπίτι με το παιδί. Επίσης, συζητούμε πώς ε, οι τοπικές ε, αυτοδιοίκησεις μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους συμβουλευτικά όργανα για να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία της ε, εκπόνησης, ανάπτυξης νέων οδηγικών θα ξεκινά από κάτω προς τα πάνω. Βεβαίω συμμερίζομαι απόλυτα την σημασία των όσων είπαν και οι προηγούμενοι για θέματα όπως η συμφιλίωση τη επαγγελματική και κοινωνική ζωή, ε, υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη. Και τώρα για πέντε λεπτά δίνουμε το λόγο καταρχήν στην ε, συνάδελφο Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν στο πολιτικό γραφείο των ΑΚΕ και προείδρευα, αλλά χρειάστηκε να έρθω εδώ, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Καταρχήν ευχαριστώ ε, για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τις ομιλήτρες και θα ήθελα να τονίσω μερικά επιμέρους σημεία και σχόλια. Βέβαια είχαμε μια συνάδελφο στην αίθουσα που όσο έλειπα κράτησε σημειώσεις και με πληροφόρησε. Όπως βλέπετε όλα είναι δυνατά για μια γυναίκα όταν θέλει. Καταρχήν χρειαζόμαστε πληροφορίες και δεδομένα ακριβή και για να διαμορφώσουμε συγκεκριμένε πολιτικές και για να υπάρχει η σωστή εποπτεία. Υπάρχει έντονη άνηση μεταχείριση βάρος των γυναικών που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θυμάμαι, είχαμε μια έκθεση με την Λίβα Γιαρόκοβα, Γιαρόκα για την κατάσταση των Ρώμα γυναικών. Αν δεν ξέρουμε για πόσα άτομα μιλάμε, είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συστή πολιτική αν δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Και μπορώ να πω ότι όλες οι συνάδελφοι στην Επιτροπή θα συμφωνήσουν ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαία. Δεύτερον, χρειαζόμαστε πόρους, ευρωπαϊκά κονδύλια για τον οδικό χάρτη. Σημαντικές οι αξίες, αλλά αξίες έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους για τον οδικό χάρτη με ευρωπαϊκά κονδύλια. Να σου πω τι συμβαίνει στην Ουγγαρία το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας δημιούργησε την ίδια ακριβώς ομάδα με τους ίδιους ακριβώς στόχους, τους έξι στόχους, τους δικού μας. Έχουμε ωραίες ιδέες και συστάσεις. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχει μέθοδος για την ίσης, ίσης αμοιβή. Χαίρομαι για το ότι μια συνάδελφος θα κάνει μια έκθεση για τις ίσες αμοιβέ. Και λέει η έκθεση αυτή, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, θα χρειαστούμε 70 χρόνια με την νομοθεσία που έχουμε για να επιφέρουμε την εξίσωση των μισθών. Αυτό είναι απαράδεκτο. Χρειαζόμαστε πίεση λοιπόν. Να υποχρεωθούν επιχειρήσει που έχουν πάντοτε 100 απασχολούμενε, να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα που να λέγεται πρόγραμμα ποιότητα. Όπου στο πρόγραμμα αυτό θα δεσμεύονται επιχειρήσει να προστατεύσουν του τροτού Απασχολούμενος ιδιαίτερα τις γυναίκες. Έστω και αν αυτό σημαίνει επιπλέον διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Μετά έχουμε άλλες στρατηγικές. 2020. Μετανάστευση. Χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το να πληρώνται οι γυναίκες λιγότερο για τη δουλειά που κάνουν και οι άντρες είναι παράνομο. Ελπίζω η Ισπανική Προεδρία να επιμείνει να αρθούν αυτές οι ανισότητες. Αλλά ακόμα και αν βάλει το θέμα στο τραπέζι της ημερήσιας διάταξης, χρειάζεται βελτίωση του δικού χάρτη. Πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες που δεν έχουν σύστημα προστασίας να εισάγουν ένα τέτοιο και να γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Και εδώ χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες που θα τις συλλέγουν οι τοπικές αρχές και τα κράτη-μέλη το παρατηρείο να λειτουργεί σωστά. Συμφωνώ το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να έχει τη διάσταση mainstreaming και αυτό. Πολλά λεφτά έχουν δοθεί για την αυτοκίνητο βιομηχανία και για τις τράπεζες. Ξέρουμε όμως ότι η οικονομική κρίση έπληξε κυρίως τους άντρες, γιατί περισσότερο άντρες ασχολούνται στους τομείς που επλήγησαν, αυτοκίνητο βιομηχανία, τράπεζες κλπ στις τράπεζες επειδή εκεί που οι γυναίκες ήταν επικεφαλής η κρίση ήταν λιγότερο έντονη πάντως οι γυναίκες είναι πολύ πιο τρωτές όσον αφορά το χώρο εργασίας σας ο άντρες μετά έχουν ε, ε, προγράμματα ε, εξόδου από την απασχόληση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και εδώ θα σταματήσω σιγά σιγά γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Κάποιος ε, είπε το κέντρο για την ισότητα των ανδρών γυναικών. Εγώ έχω ένα πρόβλημα για το EMPLG, το κέντρο που υπάρχει στην Κομισιόν για το θέμα αυτό. Αν παραμείνει στη Γενική Διεύθυνση για τις Απασχόλησεις και η Ουγγαρία θα έχει το, την επιτροπή αυτή, Καλώ τους συναδέλφους να προσέξουν αυτή την αναδιάρθρωση που θα γίνει για να μην χαθεί η ευκαιρία να υπάρξει συγκεκριμένη δράση. Και ας μην ξεχνάμε φυσικά την ενέργεια, το περιβάλλον, όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν στον οδικό χάρτη. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκουρμαή. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη τώρα. Ευχαριστώ. Οποία πρόοδος. Βλέπουμε πόσο θετικό είναι ο οδικό χάρτη. Η ισότητα των γυναικών και των ανδρών στα τα τελευταία 60 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προοδεύσει πολύ. Δικαίωμα ψήφου, υψηλά αξιώματα στι επιχειρήσει, στον τομέα τη υγεία, στα νομικά επαγγέλματα. Μέχρι και γυναίκε πιλότου, παίρνουν τις αποφάσεις για το πώς θα ζουν, έχουν έγκαια ιδιοκτησία, αποφασίζουν για την υγειονομική περίθαλψή τους. Όλοι εργάζονται σκληρά και οι γυναίκες αλλά και οι άντρες μας βοηθούν, αλλά δεν επαρκούν αυτά. Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Δεν υπάρχουν ίσοι μισθοί για τις ίδιες δουλειές δεν ε, υπάρχουν οι ίδιες εμπειρίες στο χώρο εργασίας. Ε, τα συνταξιδοτικά δικαιώματα είναι άνισα γιατί οι γυναίκες μόνο στο σπίτι να φροντίσουν τα παιδιά. Οι ανισότητες μισθολογικές διευρύνονται γιατί υπάρχει και οικογενειακή βία, υπάρχει και παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Ε, το θέμα της πολιτικής για την προστασία των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό εντάσσουμε το διάλογο μας, αλλά ε, πρέπει σε εθνικό επίπεδο να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, γιατί ποικίλει από χώρα σε χώρα και άρα πρέπει να αναρωτηθούμε προς τα που οδεύουμε. Στρατηγική της Ένωσης αυτό χρειάζεται. Ναι, αλλά χρειάζεται και εθνική στρατηγική. Και όταν μιλάμε για τις γυναίκες ε, πρέπει να εστιαζόμαστε στο εθνικό επίπεδο. Δεν γίνεται, πρέπει να προσεγγίσουμε τις γυναίκες σε τοπικό επίπεδο. Ε, ό,τι και να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται να υπάρχει στενή σχέση με την καθημερινή ζωή των γυναικών. Η δική μου πολιτική ομάδα θα πρέπει, πιστεύει ότι θα πρέπει η ηγετική θέση να έχει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σε ένα πιο προσωπικό τόνο θα έλεγα ότι το πλέον σημαντικό είναι το δικαίωμα επιλογής για τις γυναίκες. Πού πάνε, τι κάνουν, να μπορούν να διαλέγουν, πού δουλεύουν, αν θα δουλέψουν. Δηλαδή η μεγαλύτερη χειραφέτηση των γυναικών για να μπορούν να αποφασίζουν να κάνουν αυτό που επιθυμούν. Μπορώ να Είμαι ε, μια οικιακή επιστήμονας, ε, έτσι λέγεται η νοικοκυρά. Ε, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι γίνεται με τη σύνταξή τους όταν επιλέξει κάποιος να δουλεύει στο σπίτι. Ε, φαθείς ομάδες, φτώχεια, πορνεία, θύματα βίας, θύματα σωματεμπορίας. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τύχουν τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωση, να βοηθήσει η Ένωση τα κράτη-μέλη να ε, προωθήσουν αυτά τα ζητήματα, η εκπαίδευση, να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ε, είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο και λέγαμε γιατί μας αρέσει το ροζ ε, λόγω των γονιδίων μας ή έχουμε το δικαίωμα να μας αρέσει και το μπλε και το ροζ. Ε, επίσης ε, να διδάξουμε στα παιδιά ότι και στα αγόρια και στα κορίτσια ότι έχουν ίσα δικαιώματα ε, μέσα από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μέσα από τους διαφόρους φορείς που πράγουν την ισότητα πρέπει να κινηθούμε και σε ορισμένους τομείς χρειάζεται μεγαλύτερη αξιοπρέπεια για τις γυναίκες αλλά στα συνταξιδοτικά καθεστώτα τα επιδόματα για τα παιδιά παραδείγματος χαρινέμενα, αλλά μην ξεχνάτε αυτές τις στρατιές των γυναικών. Γιατί εσείς μας μιλάτε για τις υψηλές ε, θέσεις επιχειρήσεις αλλά οι στρατιές μεγάλες των γυναικών ε, χρειάζονται μια πιο βασική αξιοπρέπεια, οικονομική ανεξαρτησία, να υπάρχουν συστήματα υποστηρίξης, καλός διάλογος, ε, οργανώσεις που θα τις βοηθούν. Τώρα για την νομοθεσία ας είμαστε προσεκτικοί, ας μην υπερνομοθετούμε. Κυρία Βασιλείου, για αυτά που μας είπατε, ήθελα να ρωτήσω, να σας πω ότι ναι, πρέπει να είμαστε προορατικοί, proactive, ναι, συμφωνούμε. Ε, η βία κατά των γυναικών, μην ξεχνάμε και τη βία κατά των αντρών. Μία στις τέσσερις γυναίκε γυναίκες πέφτουν θύματα, για τους άντρες είναι ένας προ έξι. Μας πλησιάζουν για τη βία κατά των γυναικών. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Ξέρετε, οι πρόσφυγες στους καταβλισμούς προσφύγων δεν έχουν ιδέα τι κάνουμε ε, στην Ένωση. Καλύτερη ενημέρωση. Κύριε Φιλίπε, ναι, είπατε καλύτερη παιδεία, ναι, για να μπορούν να διαλέγουν, να επιλέγουν οι γυναίκε. Ε, πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τι θέλουν να κάνουν. Ε, και λέει η γυναίκα, μα εγώ με οικιακά ασχολούμαι απλώς. Μα πώς απλώς. Ε, είναι δύσκολο επάγγελμα τα οικιακά. Η τελευταία ομιλήτρια μας ε, μίλησε για την ομοθεσία για την απασχόληση. Μας τα αφήσουμε άθικτο γιατί θα πλήξουμε περαιτέρω τις γυναίκες. Πρέπει να κινηθούμε προσεκτικά αν υπερνομοθετήσουμε, ξέρετε. Δεν βοηθάτε τις γυναίκες. Οι εργοδότες κάνουν, ε, παίρνουν τις αποφάσεις που θέλουν. Έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ε, ας δούμε τι συμβαίνει πραγματικά ε, στον κόσμο. Ε, η νομοθεσία πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών για να ρυθμίσουν την κατάσταση στις χώρες τους. Κυρία Πάικ, που είσαστε εσείς. Δεσποινής είστε κυρία, δεν ξέρω, θα σας πω κυρία. γίνεται η επιλογή ότι θα παραμείνει γυναίκα στο σπίτι παρότι εργάζονται και οι δύο ε, ναι, πρέπει να σταματήσω. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η κυρία Πάικ, λοιπόν. Thanks. I'll deal in a Θα τα πάρουμε τυχαία σειρά όλα αυτά τα ζητήματα που άκουσα. Ε, μα, σας μίλησα για την μελέτη, την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Θα δημοσιευθεί σύντομα. Κάποια από τα πορίσματα δεν ξαφνιάζουν, αλλά πάλι είναι αξιόλογα διότι θα μας βοηθήσουν για να παρουσιάσουμε σωστά τις νέες πολιτικές. Τα κράτη-μέλη, ναι, έχουν ζωτικό ρόλο και οι κοινωνικοί εταίροι, όλοι οι φορείς. Ε, δεν ισχυριζόμαστε ότι με τον οδικό χάρτη, τη στρατηγική, το πλαίσιο, όπως και να το πούμε, ε, θα έχουμε την απόλυτη σοφία και την αυθεντία που θα κατεβαίνει από τις Βρυξέλλες ε, ε, και ότι θα αποτύχουν αυτοί τόπου που δεν το καταλαβαίνουν. Όχι, πρέπει να περάσουν όλα μέσα από τις δράσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα κράτη-μέλη για τους εργοδότες. Ένα πράγμα που θέλουμε να γίνει με την επόμενη πενταετία με τη στρατηγική είναι να είναι πιο απασχολήσιμοι οι γυναίκες. Υπάρχει το χάσμα ως προς το επιχειρηματικό πνεύμα, αλλά ε, θέλουμε να πληρωθεί το κενό με περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν έρθετε, είχα εξηγήσει την κατάσταση, σημειώνω τα σχόλιά σας. Θα επανέλθω στη δομή όταν περάσω στο gender mainstream για την πολλαπλή διακριτική μεταχείριση που ε, τόνισε η Λίβια Γερόκα. Βεβαίως. Θα πρέπει αυτό να αποτελεί αναπόσπαστο το κομμάτι της πολιτικής. Όλες οι πτυχές που φέρνουν επί της ισότητας, η πολλαπλή διακριτική μεταχείριση, όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καλύψουμε και άλλες ομάδες, ας το πω έτσι. Κάποιος μίλησε για το ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, τα θέματα των γυναικών για την ένταξη των ΡΟΜ, για οποιαδήποτε πολιτική απασχόληση. Έχουν γίνει πολλά για την ε, πολλαπλή διακριτική μεταχείριση και ε, κάναμε και ανακοίνωση στις 2 Ιουλίου του 2008 που είχε ενδιαφέροντα σημεία και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο της πολλαπλής διακριτικής μεταχείρισης και πώς εκφράζεται στα κράτη-μέλη και ξέρετε υπάρχουν και μη καπαόμικρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ε, ασχολούνται με ακριβώς αυτό ε, το ζήτημα, πώς δηλαδή μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα πολλαπλής διακριτικής μεταχείρισης. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που πολλές φορές χάνονται ε, για τα ε, άτομα που έχουν αλλάξει φύλλο από τον Επίτροπο Αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαμε μια σχετική δήλωση πέρσι. Υπάρχουν αυτά τα άτομα που έχουν αλλάξει φύλλο, υφίστανται σοβαρή διακριτική μεταχείριση και μπορεί αυτό να καλυφθεί από την σχετική νομοθεσία και είναι σημαντικέ οι εκθέσει των διεθνών Οργανισμού που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών είπαν ότι ε, είπε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά σε σχέση με αυτά που γίνονται για τι φυλετικέ διακριτικέ από τη μία και τις διακρίσεις κατά των γυναικών από την άλλη. Ε, στο EWL θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά ήθελα εγώ να σας υπενθυμίσω κάτι. Πέρσι έγινε μία έκθεση για την οδηγία του 2002. Ε, η Μπρι Τόμσον το ανέφερε νωρίτερα ε, και το Κοινοβούλιο ίσως θα ήθελε να τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Έχουμε και την οδηγία το 2004 για την σεξουαλική διακριτική μεταχείριση εκτός χώρου εργασίας, πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Ε, η πρώτη οδηγία που βασίζεται στο παλιό άρθρο 13. Θα κάνουμε έκθεση στο τέλος ε, του τρέχοντος έτου ε, για αυτό το θέμα, για να, την αναθεώρηση της κατάστασης, τι έχει γίνει στις ασφάλειες και στις χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε για αυτό το ζήτημα. Επίσης, οι τομείς που δεν καλύπτονται πρέπει να καλυφθούν. Η παιδεία, παραδείγματο χάρη, Οπότε σε αυτή την έκθεση θα αρχίσουμε να πραγματευόμαστε αυτά τα ζητήματα για να δούμε ακριβώς ε, ποιες θα είναι οι μελλοντικές μας κινήσεις. Σε αυτό το στάδιο δεν σας λέω ότι θα προτείνουμε νέα νομοθεσία. Αν εντοπίσουμε ανάγκη για νέα νομοθεσία θα αρχίσουμε την κανονική διαδικασία αξιολόγηση αντικτύπου και θα συνεχίσουμε Επίσης η έκθεση για την οδηγία του 2004 αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα. Για την έμφυλη βία τώρα είπαν οι διάφοροι συνάδελφοι ότι χρειάζεται ξεχωριστή οδηγία για αυτό το θέμα. Μάλιστα θα βοηθούσε αν ήσασταν λίγο πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή ακριβώς τι πρέπει να καλύπτει αυτή η οδηγία. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι το Κοινοβούλιο ε, το 2008, ε, έτσι, στη διαδικασία απαλλαγής ε, του προπολογισμού για το 2009, υπήρχε και μια προπαρασκευαστική δράση για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να εναρμονίσουμε τις εθνικές νομοθεσίες για την έμφυλη βία. Γι' αυτό το θέμα η προπαρασκευαστική δράση δρομολογήθηκε, ξεκίνησε μια μεγάλη μελέτη και θα έχουμε νεότερα αργότερα μέσα στο έτος. Νομίζω αυτό είναι ευκαιρία για να αξιολογήσουμε τα χάσματα, τα κενά που υπάρχουν και πώς θα πληρωθούν. Χρειάζεται οδηγία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βέβαια. Έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Σουηδικής Προεδρίας που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και είπαμε θα εγκριθούν στις 8 Μαρτίου. Τέλος, gender mainstreaming εντάξει των θεμάτων ισότητας φίλων ε, σε όλους τους τομεί. Ε, εμείς αναρωτιόμαστε τα ίδια με εσά. Είναι κοινή πρόκληση. Πώ ακριβώς μπορούμε να τα καταφέρουμε ούτω ώστε ε, αν και δεν ασχολούνται καθημερινά με τα θέματα ισότητας να βλέπουν τα θέματα αρμοδιότητά τους από τη δική μας προοπτική. Χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται να δούμε πώ θα εντάξουμε την ισότητα στι εξωτερικέ σχέσει, τη κοινότητα, στον τομέα τη απασχόληση πρόκειται για άτομα που δεν είναι ευαισθητοποιημένα σε αυτό το θέμα. Ε, ε, πρέπει να καταλάβουν ότι έτσι θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, θα εκπονούν καλύτερες πολιτικές, αν λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας. Ε, ε πέρα από τους ειδικού, χρειαζόμαστε και ειδικού. Ε, ε, χρειαζόμαστε δεξιότητες ως προς την ισότητα σε όλους τους τομείς όπου βγαίνουν πολιτικές. νομίζω ότι είναι μια κοινή πρόκληση για όλους και καλή τύχη στο να περάσετε αυτό το μήνυμα στους συναδέλφους σας από τις άλλες επιτροπές. Ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε στην γενική συζήτηση. Ερωτήσεις ε, από το από τα μέλη της Επιτροπής και τους παρισταμένους. Η κυρία Παβανόβα θα πάρει πρώτη το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία λόγια της κυρίας Πάικ. Προσπάθησα να καταγράψω όλες τις πολιτικές για τις οποίες θα πρέπει να είναι σημαντική η ισότητα των δύο φύλων, ε, ε, απασχόληση, αγορά εργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική βιωσιμότητα, περιβαλλοντική προστασία, στέγαση, συνθήκε διαβίωση, μετανάστευση, ένδυα, κοινωνικό αποκλεισμό, ε, καινοτομία, έρευνα, επιστήμη, μπορώ να συνεχίσω να μιλάω επάπειρον για τι πολιτικέ αυτέ, αλλά έχω την εντύπωση ότι η στρατηγική αυτή και ο, ο δικός χάρτης έχουν τη δική του ζωή, ανεξάρτητα από το τι κάνουμε εμεί εδώ και στην Ένωση και στο Κοινοβούλιο. Και σα δώσω ένα ακόμη παράδειγμα. Ενώ η Κομισιόν αποφασίζει να δημιουργήσει, ε, να ε, σε τον τομέα τη υγεία σε όλε τι πολιτικέ όλα τα κράτη-μέλη, στην αρχή τα βρήκαν δύσκολα αλλά τώρα ακολουθούν, γιατί και εμείς όπως είπε η κυρία Πάικ δεν βάζουμε την ισότητα των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές. Να είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη. Και όπως είπε και η Συνάδελφο, θα μας πάρει δεκάδες χρόνια για να καταλήξουμε σε μια πολιτική προσέγγιση βασισμένη στο φύλλο και να έχουμε ε, Ε, ίσα στατιστικά στοιχεία και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το 33 έναντι 67 γυναικών και ανδρών αντιστοίχω στην, ε, στην ε, πολιτική ζωή. Να το βάλουμε ως προϋπόθεση. Ισότητα των δύο φίλων σε όλε τι πολιτικέ, Τελεία και παύλα. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι πρόεδρο του Συμβουλίου, πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα, πρόεδρο επιτροπή, πρόεδρο ή πρωθυπουργό χώρα ή οτιδήποτε. Αυτό το περιμένουμε από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλες τις ομιλήτρες για τις παρουσιάσεις τους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. εξακολουθούν οι πολλαπλές διακρίσεις κατά των γυναικών να υπάρχουν και οξύνονται κιόλας. Η μισθολογική διαφορά πριν από πέντε χρόνια ήταν στα 15% μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και διωγγώθηκε αντί να μειωθεί. Και τώρα υπερβαίνει το 17%. Δράτω με τις ευκαιρίες παρόλα αυτά για να ρωτήσω τις ε, ομιλήτρες κάτι για το θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, της Επιτροπής μας ε, και με το οποίο εμπλέκομαι διότι είμαι η εισηγήτρια για την αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Ακούστηκε ήδη και το γνωρίζουμε όλοι ότι η συμφιλίωση ανάμεσα στην οικογενειακή προσωπική ζωή από ε, τη μία και την επαγγελματική ζωή από την άλλη είναι εκ των όνου κάνευ για την πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων. Για να επιτύχει κανείς τη συμφιλίωση αυτή απαραίτητα πρέπει να υπάρχει πλήρης επιμερισμός όλων των ευθυνών. Οικογενειακές ευθύνες, αλλά και επαγγελματικέ ευθύνε. Δηλαδή, οι άντρε και οι γυναίκε πρέπει να ζητούν την ισότητα και στην οικογενειακή και στην επαγγελματική σφαίρα. Δηλαδή, οικογενειακές ευθύνες από τη μία και αγορά εργασίας από την άλλη. Τι θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σας ως προς ε, την αξία της συμπερίληψης στην κοινοτική νομοθεσία της ε, άδεια πατρότητας. Σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχει άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας και γονική άδεια. Σε ευρωπαϊκή επίπεδο προβλέπεται μόνο άδεια μητρότητας και γονική άδεια. Είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να περάσουμε αυτό το μήνυμα για να καταπολεμήσουμε στερεότυπα που ανέφερε η κυρία Πάικ μεταξύ άλλων μιλώντας για αυτή την μελέτη όπου αναφέρεται ότι οι ίδιες οι γυναίκες πιστεύουν ότι εκείνες πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Ε, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αλλά μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα και δια της νομοθετικής οδού. Οπότε, Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Η μητρότητα και η πατρότητα κατά τη γνώμη σας δεν είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος ε, και άρα πρέπει να ε, την χάνουν ισότιμης μεταχείριση και να συμπεριληφθούν στην ίδια οδηγία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις σχετικά με τη μελλοντική πολιτική προς την Κομισιόν επίσης. Κάτι που δεν αναφέρθηκε ρητά είναι η μάχη κατά των στερεοτύπων. Ξέρουμε ότι στερεότυπα υπάρχουν ε, παντού και κατά των γυναικών φυσικά υπάρχουν. Σήμερα στην αγορά εργασία παρά την κρίση υπάρχουν ε, θέσει απασχόληση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι. σε μερικά εξειδικευμένα επαγγέλματα και σε τεχνικά. Παραδείγματο χάρη, οι ηλεκτροσυγκολητέ, ε, οι οικοδόμοι. Πολύ λίγε γυναίκε πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα. Το ίδιο ισχύει για την κατάρτιση. Στην κατάρτιση δεν γίνεται σωστά αμερόληπτα υπέρ και των δύο φίλων. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμηθούν αυτά τα στερεότυπα. Βέβαια και οι άντρε πολλέ φορέ είναι θύματα στερεοτύπων. Σπάνια βλέπουμε α πούμε νηπιαγωγού άντρε. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Στο δημοτικό δάσκαλοι υπάρχουν. Μειοψηφία βέβαια είναι. Παλιότερα ήταν η σούπερ πλειοψηφία οι δάσκαλοι νηπιαγωγοί άντρε δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Πρέπει όλα αυτά να τα απομυθοποιήσουμε με ένα είδο θετική διαφήμιση κατά κάποιο που θα, θα πρέπει να κάνουμε. Στην αρχή τη επαγγελματική μου ζωή μετά το στρατό, δεν μπορούσα να βρω δουλειά και έκανε το γραμματέα σε μια γυναίκα δικηγόρο. Ε, χτυπούσε την αλληλογραφία και λοιπά όλη την ημέρα και το βράδυ γύριζε στο σπίτι και ετοίμαζε το φαγητό. Πριν πολλά χρόνια βέβαια αυτό. Τέλο πάντων. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη μάχη αυτή κατά των στερεοτύπων. Με καμπάνια. Καμπάνια δημοσιότητε, καμπάνια μέσω του τύπου. Αμφίδρομη και για του άντρε και για τι γυναίκε. Τα στερεότυπα. Δεύτερο, η βία σε βάρος των γυναικών. Μοιραία, θυμάμαι, και στο Βέλγιο και στον Καναδά κυρίω, μια καμπάνια που αφορούσε κυρίω του άντρε. Ευαισθητοποίηση των ανδρών προ τη βία κατά των γυναικών. Υπάρχει η σωματική βία, η ηθική βία, η ψυχική βία, μην τα ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο η σωματική βία. Είναι ιδιαίτερα βία βέβαια και ομοία. Ε, μια άσπρη κορδέλα που βάζουν στι 27 Νοεμβρίου στον Καναδά ε, μια νέα κοπέλας σε ένα τεχνολογικό κάμπους στον Καναδά επαναλαμβάνω από ένα νεαρό που είπε ότι αυτό το κάμπο πρέπει να είναι μόνο για άντρε. Τι δουλειά έχει η κοπέλα εδώ και τη σκότωσε. Σκότωσε 15, 15 φοιτήτριε. Και οι άντρε ανάλαβαν να δώσουν τη μάχη. Είπαν απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά στον Καναδά. Γιατί οι άντρε δεν είναι όλοι τέρατα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση των ανδρών για την βία κατά των γυναικών και αυτό είναι μια ε, ενδιαφέρουσα προσέγγιση που δεν θα πρέπει να την ε, παραμελούμε. Πρόεδρος. Μάλιστα θα ακούσουμε τους λοιπούς συμμετέχοντες στην ακρόασή μας. Ένα λεπτό έχετε έκαστο στη διάθεσή του. Μην κάνετε δηλώσεις παρακαλώ, μόνο ερωτήσεις, έτσι. Μύρια Μπλόμπι I'm here. Hello. Um, Εγώ εκπροσωπώ το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτοδιοίκησης μέσω μιας οργάνωσης που ονομάζεται ε, Συμβούλιο για τις Ευρωπαϊκές, τους Ευρωπαϊκούς Δήμους και Κοινότητες. Θέλω απλώ να πω ότι οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ τη Ευρώπη μπλέκονται πολύ ε, σημαντικά στην εφαρμογή των δράσεων στι πόλει, στι περιφέρειες, στα συμβούλια για την πρόθεση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι απλό και σύντομο. Τα επίπεδα τα τοπικά και τα περιφερειακά θα ληφθούν υπόψη στη νέα στρατηγική που θέλετε να εκφωνήσετε και που ελπίζουμε να εφαρμόσετε και σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ανή Ελ. Χαλεβίβ. Ευχαριστώ. Σύντομο ερώτημα κι εγώ από το, την υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την, για την ισότητα των δύο φύλων. Το ερώτημά μου για την, είναι για τη διαδικασία της διαβούλευσης για τη στρατηγική. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους ε, μέσω της νομοδότησης ε, για το μέλλον του οδικού χάρτη, αλλά αναρωτιέμαι, τα κράτη-μέλη θα έχουν και άλλες ευκαιρίες να δώσουν και άλλες απόψει πριν από το τέλος του 2010. Υπάρχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ε, Άννα Καρανάβου τώρα, παρακαλώ. Ε, πρώην... Η κυρία Καραμάνου εννοεί, πρόεδρος, ε, πρώην βουλευτής, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Περιτώ να σας πω πόση χαρά νιώθω που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση για την οποία σας συγχαίρω, διότι και εγώ υπήρξα μέλος αυτής της Επιτροπής και πρόεδρος για δυόμιση χρόνια και ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ε, ερωτήσεις οι οποίες αφορούν όλο το πάνελ αλλά όλος ιδιαίτερος τη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών του οποίου λόμπι εκτιμώ πάρα πολύ την ε, δραστηριότητα. Θα κάνω τις ερωτήσεις μου στα αγγλικά για να είμαι ε, καλύτερα κατανοητή. Is there any interrelationship? Do you think that there is interrelationship between social, religious and cultural patterns of male dominance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 του... Νομίζω ότι τώρα είναι ώρα σε, μια, σε ένα, συστηματικό τρόπο πρέπει να εμπλακούν και οι άντρες σε ένα συστηματικό προγραμματισμένο τρόπο. Η ισότητα των δύο φύλων είναι υπόθεση και των αντρών, ναι ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλωσορίζουμε και πάλι στο Κοινοβούλιο σήμερα. Αν Κατρίν σιγά, τώρα, παρακαλώ. Καλημέρα. Ε, κοιτάξτε, λέμε ο τίτλος επιτροπής, ε, το όνομα της επιτροπής είναι ισότητα των φίλων και δικαιώματα των γυναικών. Γιατί δεν μιλάμε για τα, τις ευθύνες των γυναικών και τι εννοείται με τα φύλλα. Τους άντρες δεν τους έχετε ξεχάσει. Δεν σου αναφέρετε. Μήπως ε, υπάρχει διάκριση όταν μαζεύονται πολλές γυναίκες και ξεχνάμε τις διακρίσεις ανάμεσα στις γυναίκες. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Μιλάμε επίσης για πόρους που πρέπει να κινητοποιηθούν για να πληρώσουμε τα σπασμένα όταν έχει κακοποιηθεί κάποια γυναίκα, όταν είναι μόνη μέχρι να βρει καινούριο σύντροφο, για να βρει οικονομική σταθερότητα μπορούμε να κινητοποιήσουμε πόρους και για την ε, ε, ε, παιδεία, για τις γυναίκες, για τους νέους και τις νέες, για να γνωρίζουν καλύτερα την ταυτότητά τους, για να μην δημιουργούνται τα προβλήματα, να έχουν ισχυρά ερίσματα, να οικοδομούν τη ζωή τους σε μια καλή ψυχολογία και σε μια καλή ανθρωπολογική γνώση της ανθρωπότητας. Αυτό, αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται μέσα στα σχολεία. Μήπως προκύπτει το πρόβλημα επειδή δεν κατανοούμε οι μεν τους δε. Και άρα δημιουργούνται προβλήματα και στις σχέσεις, ε, προβλήματα έλλειψης κατανόησης ε, και ξέρετε τα προβλήματα αστάθειας στα ζευγάρια είναι γενικότερα ε, προβλήματα κοινωνικής αστάθειας. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, για όλες τις ερωτήσεις σας. Δείχνουν πόσο μεγάλη δέσμευση και προσήλωση έχετε για αυτά τα ζητήματα. Τώρα θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Σε τρία λεπτά έκαστη παρακαλούμε για να ακούσουμε και τη σύνοψη της εισηγήτριάς μας στη συνέχεια. Πριν δώσω το λόγο στις ομιλήτριες. Θα ήθελα να τονίσω ότι η δουλειά μας στην Επιτροπή Γυναικών είναι για να, να οικοδομήσουμε μια καλύτερη κοινωνία και για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες. Μαζί αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη κοινωνία ανεξαρτήτως φύλου να έχουμε μια ισότιμη μεταχείριση σημαντική για όλους ώστε να ζούμε όλοι σε μια κοινωνία που υπάρχει σεβασμός για το άτομο ανεξαρτήτως φύλου. Θα δώσω το λόγο τώρα στις ομιλήτριες ε, της ομάδας ε, συζητήσεων του πάνελ. Η κυρία Βασιλείου, ε, Βασιλιάδου, συγγνώμη, έχει τρία λεπτά για να απαντήσει. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, Πρόεδρε, σε τρία λεπτά. Ακούσαμε πολλά, δεν θα σχολιάσω τα πάντα. Ένα όμως από τα βασικά που, ακούστηκαν, που ακούστηκε από όλους σχεδόν ήταν η βία εναντίον των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ε, ψάχνει απαντήσεις σε σχέση με τη νομική βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό. Ε, σε αντίθεση με κάποιον από τους συναδέλφους που δυστυχώς έφυγε και που λέει εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε ε, την νομοθεσία η οποία μπορεί να αλλάξει τις νοοτροπίες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν όταν φτάνουμε στο επίπεδο ευρωπαϊκών στρατηγικών η Κομισιόν να λάβει συγκεκριμένη απόλυτη θέση και να πει ότι η Ευρώπη το θέλει αυτό. Όταν ερχόμαστε στο επίπεδο των κρατών μελών έχουμε κράτη-μέλη που υπογράφουν το ΣΥΝΤΑΝ και όταν υπογράφουν ε, εντάξει αλλά όταν πάμε να εφαρμόσουν το ΣΥΝΤΑΝ δεν γίνεται τίποτα. Είναι λοιπόν θέμα που πρέπει να το βλέπουμε από καιρού καιρών. Ο λόγος για τον οποίο τώρα χρειαζόμαστε τα δεδομένα και τα στατιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ακριβώς επειδή μπορούμε να καταλήξουμε σε οποιοδήποτε ε, νούμερο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε μία στις έξι γυναίκες ε, πέφτει θύμα ξυλοδαρμού ή μπορούμε να πούμε ότι δαπανουνται τόσα δισεκατομμύρια στην ε, Ευρώπη. Είναι αυτό το κόστος ας πούμε της βίας που στην οποία υποκειται οι γυναίκες. 35 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. 35 δισεκατομμύρια ανά την Ευρώπη. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και σαφή. Η βία λοιπόν και η θέση μας εναντίον της βίας είναι πολύ σαφής. Μιλούμε για βία εναντίον των γυναικών, κυρίως μιλούμε για τη βία των αντρών εναντίον των γυναικών και αυτό προσπαθεί να επιτύχει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Είναι θέμα δομών. Επίσης μας συζητήθηκαν κάποιες απαντήσεις για την μητρότητα, για την πρόταση οδηγίας που υπάρχει. Πρέπει να πω πως ε, η κυρία Στρέλα είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα αυτής της οδηγίας και εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα γιατί ζητούμε την, ε, να συμπεριληφθούν αυτά που προτείνει η κυρία Στρέλα ε, στην πρόταση να γίνεται δηλαδή πλήρης αποπληρωμή του μισθού κατά τη διάρκεια της, μητρικής, της αδείας μητρότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα την πατρότητα και την άδεια πατρότητα, πρέπει να πω ότι α, οι απόψει εκεί δίστανται. Όχι γιατί δεν είναι απόλυτα σημαντικό. Φυσικά είναι σημαντικό και τον υποστηρίζουμε την κυρία Στρέλα που το τονίζει. Αλλά θα θέλαμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να πούμε γιατί δεν έχουμε μία πρόταση για την πατρότητα. Υποστηρίζουμε αυτά που λέει η κυρία Στρέλα. Αλλά δεν έχουμε δει και καμία άλλη εναλλακτική πέραν, αυτή, τη ε, πέραν αυτής της πρότασης. δεν λέμε ότι η άδεια πατρότητα θα πρέπει να εμπίπτει στην, πρόταση για την ε, άδεια μητρότητα. Θα μπορούσε να υπάρξει μια ξεχωριστή ε, πρόταση γι' αυτό. Ε, αυτά θα σταματήσω εδώ γιατί και χρόνο δεν έχουμε και τα ερωτήματα ήταν πάρα πολλά. Ελπίζω να απάντησα. Μάλιστα, τώρα η κυρία Φιλίπε παρακαλώ. Ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έρχεται από την ε, κυρία Εστρέλα και έχει ιδιαίτερη σχέση με την Πορτογαλία. Στη χώρα μου έχουμε προς το παρόν 20 ημέρες προβλέπονται για την άδεια Αλλά δεν τις ε, χρησιμοποίησαν στην αρχή οι άντρες θα πρέπει, γι' αυτό σας έλεγα ότι πρέπει να επενδύσουμε στην αλλαγή νοοτροπίας ε, για να γνωρίζουν όλοι τα δικαιώματά τους και οι άντρες ε, ούτως ώστε να μπορούν ε, και οι άντρες να συμφιλιώνουν την οικογενειακή και την επαγγελματική τους ζωή και να περνάνε χρόνο με τα παιδιά τους. 50% των αντρών τελικά αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διάταξη και για τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να, γίνεται, ε, να ασκείται αυτό το δικαίωμα και για να καταργηθεί διακριτική μεταχείριση μέσα στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα αγωνιστούν και οι άντρες και οι γυναίκες ε, για να επιτύχουμε το στόχο μας. Τώρα κάτι άλλο. Μίλησαν πολύ για τους μισθούς και για την ισότητα τη μισθολογική. Μα δεν είναι αυτό το βασικότερό μας πρόβλημα στην Πορτογαλία. Είναι η ίσια αξία ε, το, της εργασίας. Ε, δηλαδή ε, υπάρχουν τομείς όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ή όπου γενικότερα υπάρχουν χαμηλότεροι μισθοί. Άρα θα πρέπει να γίνει σωστή ανάλωση για την οργάνωση της αγοράς εργασίας ούτως ώστε να αναγνωριστεί η αξία της εργασίας γιατί η εργασία δεν έχει φύλλο και εν πάση περιπτώσει να αμείβεται σωστά η αξία οποιασδήποτε εργασίας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι γιατί είναι ε, πιο σημαντικό το πρόβλημα. Τι να σας πω, να συγκρίνω ε, το ράφτι με τη μοδίστρα. Μπορώ παραδείγματο χάρη να συγκρίνω δύο μηχανικούς που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και δεν παίρνουν τον ίδιο μισθό, την ίδια ε, μηχανή χρησιμοποιούν. Και πέρα από την ισότητα στην εργασία και την ισότητα των μισθών, πιο σημαντικό είναι να αξιολογούνται ε, σωστά ε, οι εργασίες, οι θέσεις εργασίας. Ε, παραδείγματος χάρη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ξέρετε πόσα πληρώνται μέσα στα εργοστάσια αυτοί που είναι στις αλυσίδες συναρμολόγησης των αυτοκινήτων. Πολύ χαμηλούς μισθούς έχουν σε σχέση με άλλα αντίστοιχα επαγγέλματα. Πρέπει να κατοχυρώσουμε τις ίσες ευκαιρίες όχι μόνο για τη δουλειά αλλά και για την κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση και πρέπει να καταλάβουν ναι, όλοι ότι είναι κοινό αγώνας, κοινό μέτωπο και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καϊβανόβα τώρα. Въпросите са много интересни, както и... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα ετέθησαν και η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε δύο θέματα. Καταρχήν, γονική άδεια. Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τον όρο άδεια ε, μητρότητας με τον όρο γονική άδεια. Γιατί όταν μιλούμε για άδεια μητρότητας, αυτό συνήθως σημαίνει δικαίωμα και υποχρέωση της μητέρας. Αν αντικαταστήσουμε το, ε, όρο, τον όρο μητρότητα από το γονική άδεια, ε, με το γονική άδεια, ίσως να σπάσει το στερεότυπο αυτό. Ίσως αυτό δηλαδή να έχει και λίγο ψυχολογικές επιπτώσεις ώστε να γεβερεθεί το, το χάσμα μεταξύ της διαφορετικής μεταχείρισης που υπάρχει για τους άντρες και τις γυναίκες. Η συνάδελφη από την, ε, η από την Πορτογαλία μίλησε για την ε, αύξηση των ημερών άδεια. Είναι μια καλή αρχή αυτό. Ας βασιστούμε σε αυτό και ας συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσει έναντι των εργοδοτών που έχουν πάνω από 50 εργαζόμενους, να προετοιμάζουν δηλαδή ένα πλάνο ετήσιο για τις ίσες ευκαιρίες. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και έναν ετήσιο έλεγχο, μια ετήσια εποπτεία για τις διατάξεις που διέπουν την ε, ίση μισθολογική αμοιβή. Τώρα, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επίσης έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Θα πρέπει οι προσπάθειες αυτές να επικεντρωθούν στο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να την χάνουν ίσης μεταχείρισης και να ξεριζώσουν τις ανισότητες. Αυτό μπορεί να το καλύψει και η εργασία του Κοινοβουλίου, αλλά και η νέα, να καλυφθεί και στα πλαίσια της νέας οδηγίας. Ευχαριστώ. Και, ε, Mrs. Η κυρία Πάικ ε, θα πάρει το λόγο τώρα γιατί της απίφθηναν ε, διάφορα ερωτήματα οι συμμετέχοντες. Yeah μερικά σχόλια. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πολιτικές που πρέπει να έχουν μια διάσταση φύλου, ισότητας των φύλων. Ήδη σε έναν βαθμό υπάρχει υποχρέωση μας να το κάνουμε διότι η νέα συνθήκη και η παλιά συνθήκη δημιουργεί την υποχρέωση την Ένωση να άρει τις διαφορές και να προωθεί την ισότητα. Δυστυχώς αυτό δεν αρκεί. Είναι βάση όμως σημαντική για το mainstreaming ως προς τα φύλλα. Πιο ισχυρή βάση τώρα σε σχέση με άλλου είδους άγγιση μεταχείριση του νέου άρθρο 8 δηλαδή της συνθήκης πρέπει να το δούμε παράλληλα με το άρθρο 10. Πάντως το 8 είναι ε, το ατού προκειμένου η Ένωση να προωθήσει την ισότητα. Τώρα για το σχόλιο για το Ηνωμένο Βασίλειο και το input όσον αφορά τη στρατηγική. Το συζητήσαμε πολύ με τις κυβερνήσεις, κάναμε μια διάσκεψη εδώ, ήρθε ο Βρετανός Υπουργός, μίλησε στο υψηλό επίπεδο ομάδα για το mainstreaming, το οποίο εκπροσωπώ, το συζητήσαμε. Ενδιαφέρουσα συζήτηση και στο Συμβούλιο στις 13 Νοεμβρίου τα φύλλα και η οικονομική ανάπτυξη όλες οι κυβερνήσεις είπαν τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για την ισότητα των φύλων. Όλα αυτά βέβαια τα στοιχεία θα μας βοηθήσουν να επεξεργαστούμε τη στρατηγική μας, αλλά το Μένο Βασίλειο και οι άλλες κυβερνήσεις θα έχουν την ευκαιρία από τη στιγμή που θα υποβάλει η Κομισιόν το σχέδιό της για τα επόμενα πέντε χρόνια να έχουμε ένα εταίρο στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο προκειμένου να εφαρμοστούν όλα αυτά γιατί μπορούμε να λέμε εσείς και εμείς πράγματα αλλά αν δεν τα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη δεν σημαίνουν τίποτα. Έχουμε λοιπόν input από τις χώρες αλλά από τη στιγμή που θα επεξεργαστούμε και θα υποβάλουμε τη στρατηγική θέλουμε οι χώρε μέλη να φροντίσουν να γίνει η δουλειά και για την ισότητα των φίλων και για όλες τις άλλες πολιτικές που συζητάνε οι κυβερνήσει τη Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στην συγγήτρια μας, συγγνώμη τώρα, στην κυρία Φίγκη Ρέιντο για να προσπαθήσει να συνοψίσει αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που τώρα ολοκληρώνεται ε, και να μας μιλήσει για τις, ε, τα νέα στοιχεία που ε, προέκυψαν από τις παρεμβάσεις όλων των βαρεσταμένων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχετε δίκιο. Ε, μόλις ολοκληρώνεται μια πολύ σημαντική συζήτηση, μια ακρόαση που κατά τη γνώμη μου άγγιξε όλες τις συνιστώσεις της ζωής των γυναικών και της κοινωνίας γενικότερα. Γιατί, ξέρετε, είναι θεμελιώδης κομμάτι της κοινωνίας οι γυναίκες και είναι και η πολυπληθέστερη ομάδα εξετάσαμε τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να βελτιώσουμε την κοινωνία. Για να βελτιωθεί η κοινωνία πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί η ζωή των γυναικών. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σεβασμός της αξιοπρέπειας ε, των γυναικών ε, ε, όπως όλων των ανθρωπίνων όντων ε, να κατοχυρώσουμε, να περιφρουρήσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα που διέπνευσε ολόκληρη τη συζήτηση, κυρίως το πρώτο τμήμα της ακρόασης και θα ήθελα να το τονίσω και εγώ, διότι η κοινωνική ένταξη είναι ένα ζήτημα καθοριστική σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, σοβαρότατες επιπτώσεις ε, που αναφέρθηκαν προηγουμένως ε, της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που όλοι έχουμε βιώσει. Οι συνέπειες επηρεάζουν πολύ σημαντικότερα τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες οι γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις οι μετανάστριες, οι Ρώμ, οι γυναίκες που μένουν μόνες, οι ηλικιωμένες γυναίκες. μονογονεϊκές οικογένειες, έτσι λέμε, αυτό τον όρο χρησιμοποιούμε, που γυναίκες μόνες με τα που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Πολλαπλές διακρίσεις, όλες αναφέρθηκαν, γυναίκες με αναπηρίες. Δεν θα παριθμίσω τώρα όλες ε, τις ε, πτυχές του ζητήματος, αλλά όλοι γνωρίζουν πώς πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι διακρίσεις, επέφτουν θύματα διαφόρων καταστάσεων οι γυναίκες και επιδεινώνεται η κατάσταση στην Ένωση και σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Το ακούσαμε και αυτό. Οπότε, για όλες αυτές τις γυναίκες οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, να κατοχυρώσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε μιλάμε για εισοδήματα, είτε μιλάμε για εργασία, η αξία της οποίας πρέπει να αναγνωρίζεται κατά το δέον, γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζεται η οικονομική τους ανεξαρτησία ή οι τρόποι παρέμβασης για να γίνει περιφρούρηση των δικαιωμάτων γιατί χρειάζονται αυτή την υποστήριξη οι γυναίκες. Δεν ομιλούμε μόνο για την προστασία των μισθών. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που επιτρέπουν στις γυναίκες να αποτινάξουν αυτή την εξάρτηση από την οποία υποφέρουν ε, εκπαίδευση, παιδεία κατάρτιση, μορφές κοινωνικής στήριξης υποστήριξη της οικογένειας, ε, βοήθεια για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, α, και τα ζητήματα υγείας. Ε, είναι πολυδιάστατα αυτά τα ζητήματα, έτσι, σεξουαλική υγεία, αναπαραγωγική υγεία, υγεία για τις ηλικιωμένες ε, γυναίκες, συνοδευτικά μέτρα που είναι απαραίτητα. Σε μια κατάσταση κρίσης φυσικά αυξάνονται οι διακρίσεις. Αναφέρθηκε αυτό. Μεταξύ άλλων και ως προς τους μισθούς. Αυξάνονται, διωγγώνονται οι διακρίσεις. Η ένδια, αυτός ναι, ο τομέα των μεγαλύτερων διακρίσεων. Δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε σε ένα κατώτατο εισόδημα για να ζει ε, σε συνθήκες αξιοπρέπειας ε, η γυναίκα. Ε, η φτώχεια έχει γυναικείο πρόσωπο, καταδεικνύεται αυτό από τα στατιστικά δεδομένα. Πάντως, είναι σημαντικό να πάμε επί τόπου να μιλήσουμε με τις γυναίκες, να δούμε συγκεκριμένα τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη. Ε, το τοπικό επίπεδο, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιφερειακές αρχές, ε, ε, τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη γενικότερα, να έρθουμε σε επαφή και να ακούμε τις γυναίκες. Αλλά δεν φτάνει αυτό, χρειαζόμαστε και δείκτες που με κάποιο τρόπο θα μας δείξουν, θα μας περιγράψουν την κατάσταση. Οπότε θα πρέπει να ε, επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα ως προς τους δείκτες που απηχούν πίστα την πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής και σε όλες τις πολιτικές αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτατα στις γυναίκες σε σχέση με το παρελθόν σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο και εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές. Ε, αλλά ας μην ε, μεν όλα αυτά ε, ε να κινητοποιηθούμε όλοι για να το επιτύχουμε. Αναφέρθηκαν διάφορα νομοθετικά εργαλεία που θα λειτουργήσουν ως βοηθητικά εργαλεία. Στην Επιτροπή μας Συζητήσαμε σχάτως το θέμα της άδειας ε, μητρότητος και ισχυριζόμαστε ότι χρειάζεται ως αντιστάθμισμα και η άδεια πατρότητας. Δεν προβλέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχει σχετική εθνική εμπειρία. Πορτογαλία, παραδείγματος, χαρακούσαμε το παράδειγμα. Υπάρχει αυτή η θετική πτυχή που αγγίζει και τους άντρες και τις γυναίκες και καταπολεμά την διακριτική μεταχείριση και συμβάλλει και στην ανατροφή των παιδιών. Κερδίζουν και τα παιδιά από αυτό. Μην το ξεχνάμε. Ε, Αυξημένε γνώσεις της εθνική εμπειρία, ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών και διάδοση των θετικών εμπειριών. Ε, να άλλοι τρόποι με τους οποίους ε, μπορεί να δράσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να ελπίζουμε σε μια ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διάδοση των εθνικών εμπειριών. Επίσης, βελτίωση της ευιστάμενης νομοθεσίας, ε, τροποποίηση και βελτίωση της ευιστάμενης νομοθεσίας. Αυτό το ε, στον τοπέα αυτή τη οδηγία ε, που αναφέρατε μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Θα συνεχίσουμε ε, επίσης οι συνέπειες της φτώχειας, της σώματεμπορίας, ε, ε, εμπόριο ανθρώπων, κυρίως γυναικών, πορνεία, είναι όλα αυτά κατάλοιπα της κρίσης. Τα στερεότυπα, οι κοινοτοπίες που ακούμε για τους άντρες και για τις γυναίκες Όλοι αυτοί θα είναι οι στόχοι μας. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Προετοιμάζουμε τώρα το σχέδιο έκθεση που θα συνεχίσει να συζητείτε. Μπορείτε να συμβάλλετε κι εσείς με διάφορους τρόπους. Ήδη καταγράψαμε ε, τις θέσεις που καταθέσατε, τις απόψεις σας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί ε, και στην Επιτροπή με συμμετοχή των βουλευτών των διαφόρων πολιτικών ομάδων με απότερο στόχο την πρόοδο προς μια πιο δίκαιη κοινωνία για μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, αλλά σημειώνοντας κοινωνική πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση εις βάρος καν ενός ε, κοινωνική πρόοδος όπου θα εντάσσονται όλα τα, όλοι οι άνθρωποι καλύτερα και όπου όλοι θα ζούμε καλύτερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, κυρία Φιγκυρέντο και καλή τύχη με την, το σχέδιο της έκθεσης πρωτοβουλίας που έχετε αναλάβει. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Φιγκυρέντο. Δηλαδή, ε, όλοι μπορούν να συμβάλλουν για να έχουμε μια καλύτερη στρατηγική ισότητα ε, από τους ρόλους που διαδραματίζουμε καθημερινά, χρησιμοποιώντας τις δικές μας εμπειρίες και τις δικές μας γνώσεις, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε. Χρειαζόμαστε τη συμβολή όλων με κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς ε, που ε, ασχολούνται με το θέμα της ισότητας από διάφορες πλευρές ε, μπορούν να συμβάλλουν στέλνοντας θέσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Κλείνοντας να αποχαιρετήσω τις ομιλήτριες των δύο πάνε, των δύο ομάδων που ε, με τις ε, παρεμβάσεις τους ήδη συνέβαλαν πολύ στις εργασίες μας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους, ευχαριστώ όλους τους παρισταμένους και η Πρόεδρος ευγενικά ευχαριστεί και εμάς τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς.